Buenos días. Bonjour. Bonjour à tous. À toutes. Good morning everybody. Καλημέρα σας όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. We should get started. Of course, welcoming everybody around and honored and happy. Σας καλωσορίζω. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή να καλωσορίζω ξανά την Διακοινοβουλευτική Επιτροπή, 38 βουλευτές από 26 εθνικά κοινοβούλια από 19 χώρες ε, και μία υποψήφια και από μία χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έχουμε δηλαδή εξαιρετική ένδειξη του ενδιαφέροντος των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα θέματα που θα μας αποσχολήσουν σήμερα δηλαδή το που βρισκόμαστε σε σχέση με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, σε σχέση με την ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από τη θέση ενισχύ της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Θα δούμε τα σχετικά άρθρα, το 70 και 71 της Συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80, 81, 82 και 83 που αφορούν ε, την συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων όσον αφορά τον ε, χώρο ελευθερίας και ασφάλειας. Η ανταλλαγή λοιπόν απόψεων μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να αναπτυχθεί ακριβώς αυτός ο χώρος ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης με τρόπο συνεπή, συνεκτικό και με δημοκρατικό έλεγχο. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μιλάμε, όταν μιλάμε για τα εθνικά κοινοβούλια, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τους ε, πολίτες ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο είναι άμεσα ερετό και αυτό έχει την ε, σημασία του. Γι' αυτό κάθε έξι μήνες μαζευόμαστε και έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση για να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα της Οκχόλμης. Έχουμε τώρα τον ε, κύριο David Stanton, ο οποίος είναι πρόεδρος της, της Επιτροπής για θέματα δικαιοσύνης άμυνας και ισότητας της Ελλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων, που θα ε, α, έκανε την πρώτη παρέμβαση, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε ξεκινάμε εμείς με το πρώτο τμήμα της ε, συζήτησής μας. Θα εξετάσουμε την αστυνομική συνεργασία, καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις γίνονται όλο και πιο διεθνείς. Μιλάμε για σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα όταν εξετάζουμε το τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου ειδικά στην Επιτροπή μας και οι εθνικές διοκτικές αρχές πρέπει άρα να έχουν όλο και πιο στενή συνεργασία με τους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών όπως το PRUM και το σύστημα πληροφοριών Schengen και να μοιράζονται πληροφορίες, πόρους και σε κεντρικό επίπεδο της Ευρωπόλ και στο εθνικό επίπεδο. Και βεβαίως αυτό γύρει πολλά ερωτήματα για το πώς τα εθνικά και, ευρωπαϊκά, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να διασφαλίσουν την εποπτεία για να διασφαλίσουν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και κυρίω βεβαίω ε, την ιδιωτική ζωή του, όπω είδαμε τι τελευταίε μέρε. Οπότε βλέπουμε πω υπάρχει αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο πρέπει από την άλλη πλευρά να οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία ημών, εδώ εντός αίθουσα. και άρα θα δούμε συγκεκριμένα την πρόταση που υιοθετήθηκε το Μάρτιο από την Κομισιόν για την ενίσχυση της Ευρωπόλ. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα ο κύριος ε, Δίας Δεμέρα και του δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωβουλευτές. Θέλω να απευθύνω ιδιαίτερα ένα χαιρετισμό στην Βερονίκη Ματιέ που είναι η συντονίστρια μας, η Κορνίλια Evans, η οποία είναι ισχυώδης εισηγήτρια όσον αφορά το, την έκθεση για τον κανονισμό της Europol. Ιδιαίτερος με χαροποιεί το ότι βλέπω εκπροσώπους από τα 26 εθνικά κοινοβούλια, από τα 19 κράτη-μέλη. Έχω αναλάβει την εισήγηση για τον κανονισμό της Europol και του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της ε, Europol συγκροτήθηκε στις 26 Εβδόμου του 1995. Αυτό γίνεται με κάποια σύμβαση δυνάμει της συνθήκης του Μάστεχτ. Αυτό για να βελτιωθεί η λειτουργία της Europol. Κάναμε τρία πρωτόκολλα από το 2000 μέχρι το 2003. Αυτά τα πρωτόκολλα που γνωρίζετε στις 29 Τρίτου και 18 Τετάρτου του 2007 ετέθησαν σε ισχύ. Επρόκειτο για μακρά και περίπλοκη διαδικασία. Θα έπρεπε να υπάρχει πιο αποτελεσματικό ε, ούτως πιν καταστατικό για την Γεροπολό τόσο ώστε να μπορεί πιο αποτελεσματικά να καταπολεμήσει το έγκλημα. Το έγκλημα το οποίο όλο ένα και πιο παγκοσμιοποιημένο καθίσταται και με την θέση σε ισχύ της συνθήκης του Άμστερνταμ πρόκειται να αναδιοργανωθεί η Europol και να γίνει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία να έχει κοινοτικό προπολογισμό. Και γι' αυτό το λόγο στις 6 Τετάρτου του 2009 το Συμβούλιο ενέκρινε τη σχετική απόφαση αυτήν την οποία σας προανέφερα και έτσι συγκροτήθηκε αυτή η υπηρεσία του, Ευρωπαϊκού Γραφείου Γραφείο ε, Αστυνομίας δυνάμει της συνθήκης της Europol και στην, την πρώτη 12 του 2009 τέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας οπότε αυτό οδήγησε στο ότι μπορεί να υπάρχει η συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δε το άρθρο 88 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ορίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με έναν κανονισμό θα ρυθμίσουν την δομή και τη λειτουργία αλλά και τις αρμοδιότητες της Europol. Έτσι έχουν σήμερα τα πράγματα. Οπότε η Europol τώρα θα πρέπει να υποστηρίζει τις ε, εθνικές διευθυντικές ε, ε, αρχές, να τις συντονίζει κατά της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος. Επίσης, συντονίζει λοιπόν γενικότερα τις αντίστοιχε αρχές, γίνονται οι εγκληματολογικές αναλύσεις, βοηθάται γενικά η εθνική αστυνομία. Και επίσης διευκολύνονται οι διασυνοριακές έρευνες. Έχουμε τώρα ε, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να τα έχετε υπόψη ότι η πρόταση κανονισμού από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπής έγινε στις 7 Μαΐου και ακριβώς όπως υπήρχε δέσμευση χθες κατετέθη η δική μου εναλλακτική νομοθετική πρόταση. Αυτή η πρόταση ξεκινά με κάποια μεγάλη επιλογική έκθεση. Έχουμε δε 130 τροπολογίες για τη Επιτροπής στις 18 Ιουνίου έχουμε την επίσημη παρουσίαση του σχεδίου κειμένου μου ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στις 9 Ιουλίου 14, 14 κεφάλαια και 79 άρθρα διατάξεις. Με συγκεκριτές επομένως είμαι εγώ. Ε, αλλά εκτό τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχουμε τέσσερι αρμόδιε επιτροπέ ε, προπολογισμού, ελέγχου προπολογισμού, απασχόληση αλλά και των συνταγματικών υποθέσεων. Αυτό το σχέδιο εικονισμού προσφέρει πάρα πολλέ σημαντικέ καινοτομίε. Πολλέ εξ αυτών, όπω προανέφερα, θα υποστούν κάποιε αλλαγέ μέσω των τροπολογιών μου. Πρώτα-πρώτα, κάτι το οποίο θέλω να σα θέσω υπόψη, είναι το ότι καταρχήν δεν συμφωνώ με την συγχώνευση Θεπόλ και Ευρωπόλ, όπως προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτή τη συγχώνευση, επομένως, ε, θέλουν να προχωρήσουν και εγώ δεν συμφωνώ. Επίσης έχουμε και την πρόταση για την Εκτελεστική Επιτροπή που εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό θα αποδώσει, δεν θα είναι κάτι το λειτουργικό, το επιχειρησιακό. Εγώ νομίζω ότι θα αποτελέσει μια, μια υπηρεσία μέσα στη Europol που δεν θα εξυπηρετεί. Επίσης, έχουμε μια σειρά τροπολογιών και αυτό έγινε βεβαίω με την ανοιχτή με τη βοήθεια του κ. Χάστιν, ο οποίος εδώ είναι ε, εδώ στο, στο, στο Προεδρείο, που είναι ο επόπτης των ε, δεδομένων στο επίπεδο ευρωπαϊκό και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο των εθνικών μονάδων σαν σημεία επαφή με την Europol. Επίσης, κάτι το οποίο επίσης θα σας ενδιαφέρει, έχουμε καταρτήσει μία συνταγή ούτως υπήρ για το πώς, πώς θα γίνεται ο έλεγχος και η υποπτία από πλευράς Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ακριβώ όπως λέει η υπόμενη της ε, τη Λισαβόνα, είπαμε ότι θα πρέπει ε, η Europol να υπόκειται στον έλεγχο των δημοκρατικά κλεγμένων εκπροσώπων ε, των Ευρωπαίων. Και ο κοινοβουλευτικός έλεγχο που προβλέπεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα προβλέπεται ρητός εις το κεφάλαιο 9 του κανονισμού. Όμως, έχουμε πάρα πολλές μνήες σε αυτόν τον έλεγχο ε, που διαπνέουν όλο το σώμα του κανονισμού. Ο δε μηχανισμός της εποπτείας το, της Europol από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κάτι το οποίο εγώ το περιέλαβα στη δική μου αναλεκτική νομοθετική πρόταση και αυτός ο έλεγχος θα γίνεται μέσω μιας ομάδας ε, ευρωβουλευτών του βουλευτών του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού και θα, θα πρόκειται για αυτή την ομάδα αναφορά και θα προέρχονται αυτοί από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, δηλαδή την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και εκεί θα συμμετέχει και ένα ε, ένας βουλευτής από την αντίστοιχη Επιτροπή Εθνικού Κοινοβουλίου. Με αυτή επομένω τη δομή θα διαμορφώνεται, θα συγκροτείται μια τέτοια ομάδα ελέγχου από εδώ, από, την Επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου. Ξεκινάει λοιπόν από τον πρόεδρο της, της Αρμοδίας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συμπροεδρεύεται από τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και από τον εκπρόσωπο του Εθνικού Κοινοβουλίου, του κράτους μέλους που κάθε φορά θα ασκεί την Προεδρία. Οπότε και εξασφαλίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο την ε, σύνδεση, την επαφή Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα, να σας εξηγήσω ποιες θα είναι ακριβώς οι αρμοδιότητες αυτής της ομάδας, της ελεγκτικής. Θα συζητεί την ετησία έκθεση των δραστηριοτήτων της Europol. Θα υπάρχει το ετήσιο αλλά και το πολιτές πρόγραμμα δραστηριοτήτων η ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασία Δεδομένων όσον αφορά τι εποπτικέ δραστηριότητε τη Europol. Θα έχουμε την έκθεση επίση αξιολόγηση που θα κάνει κάθε πέντε χρόνια η Επιτροπή, ούτω ώστε να αναλύει την αποτελεσματικότητα του έργου τη Europol και επίση αυτή η ελεγκτική ομάδα θα μπορεί με δική τη πρωτοβουλία να καλεί ενώπιόν τη τον υποψήφιο διευθυντή της Europol, ούτως ώστε να προβαίνει βέβαια σε κάποια δήλωση και εισήγηση, αλλά και να γίνεται συζήτηση πάνω στο έργο το οποίο θα αναλάβει. Ενώπιον λοιπόν αυτή τη κοινοβουλευτική ε, ομάδα ελέγχου, επίση θα εμφανίζονται ο πρόεδρο του Διευθυντικού Συμβουλίου, ο εκτελεστικό διευθυντή, ο Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων και πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. προστασία δεδομένων επομένω από πλευρά τη αστυνομία, αλλά, αλλά θα συμμετέχει εκεί σε πολύ τακτά διαστήματα και ο Ευρωπαίο Επόπτης. Όπως είπαμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρχεται να με αυτή την ελεγκτική ομάδα, οπότε το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλιο επίσης πρόκειται να αναλύουν απειλές, στρατηγικές ε, αναλύσεις, γενικές εκθέσεις σε σχέση με τους στόχους της Europol. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητέ πρόεδρε, δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε τη βασική λειτουργία. του Κοινοβουλίου, που είναι η μεσονομική. Οπότε πρόκειται να έχουμε το σχέδιο του προπολογισμού, τις προβλέψεις, την οικονομική κατάσταση, την μεσονομική κατάσταση, οπότε και αυτή η ομάδα πρόκειται επίσης να ορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και θα ε, συζητείτε και θα κρίνετε επίσης ε, ο προϋπολογισμός της Europol. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ευχαριστώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ κύριε Δίας Ντεμέρα. Είναι σαφής η κατάσταση η πρωινή συνεδρίαση θα ασχοληθεί στην πρωινή συνεδρίαση θα, ασχοληθούμε με δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις. Με αυτό θα απασχοληθούμε όλο το πρωί και εν συνεχεία το απόγευμα θα μιλήσουμε για τη δικαστική συνεργασία. Και τέλος θα ακούσουμε κάποιες σκέψεις για την ε, ευρωπαϊκή κουλτούρα ε, συνεργασία στο δικαστικό τομέα. Αλλά ας επικεντρωθούμε καταρχήν σε αυτό το θέμα, αστυνομική συνεργασία. Και θα δώσουμε το λόγο στον Λόρδο Χάνι Οφτσίστη, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εν συνεχεία, ο κύριος Πίτερ Χάστινγκς, που είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και είναι ένας τακτικός επισκέπτης της ΛΥΜΠΕ, και των ε, διαλόγων που έχουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λόρδα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους ενός ε, Εθνικού Κοινοβουλίου ε, σε αυτή τη συζήτηση για την Europol. Μου αρέσουν αυτές οι συναντήσεις υπό την Προεδρία σας, γιατί πιστεύω ότι στον τομέα αυτό όπου κάποιες αρμοδιότητες έχουν χορηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλές ακόμα αρμοδιότητες παραμένουν στα εθνικά κράτη και θα παραμείνουν σε αυτόν τον τομέα της ε, αστυνομίας και αστυνομικής δικαστικής συνεργασίας σε ποινικέ υποθέσεις είναι πολύ σημαντικό η εποπτεία των εθνικών ε, κοινοβουλίων που ασκείται σε εθνικό επίπεδο να γίνεται ε, και να λαμβάνει υπόψη στην εποπτεία που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί αν αυτά τα πράγματα τα διαχωρίσουμε εντελώ, τότε θα τα μπερδέψουμε τελείω. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε πριν από λίγα χρόνια να διοργανώνετε αυτές τις ε, τακτικές συναντήσεις ε, και να τις πλαισιώσετε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Η Επιτροπή της οποίας προεδρεύω είχε πολλές ευκαιρίες να εξετάσει τη δουλειά και το έργο της Europol ε, στα πλαίσια πρόσφατων ερευνών που κάναμε και που δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα τους. Κοιτάξαμε την θέση της Europol στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ρόλο της στο ξέπλυμα του χρήματος και το ρόλο της στο λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, καθώς και στο κυβερνοέγκλημα. Και είδαμε πολλά από αυτά που είχε κάνει η Europol τα πρόσφατα χρόνια. Σε αυτές τις έρευνες που κάναμε και για τις οποίες δημοσιεύσαμε εκθέσεις, πραγματικά φτάσαμε ε, στην... Αξιολογήσαμε και θαυμάσαμε το έργο της ε, Europol. Γίνεται ανάλυση Γίνονται κοινέ έρευνες, ομάδες, κοινές ομάδες έρευνας για να διερευνηθούν διάφορα εγκλήματα και ο σκοπός είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος να υποβοηθηθούν ακριβώς από τη Europol. Το σοβαρό έγκλημα γίνεται όλο και πιο διεθνές. Και καθώ θα γίνεται όλο και πιο διεθνέ και καθώ οι εγκληματίες ε, υποφελούνται από τις ελευθερίες της ε, αγορά, αγοράς, ε, ακόμα και ένα νησιωτικό κράτο όπω το δικό μου να γνωρίζει ότι η εσωτερική μα ασφάλεια δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στα χωρικά μας ύδατα. Και αυτό εξηγεί το θερμό καλωσόρισμα που επιφυλάξαμε στην πρόταση που συζητάμε σήμερα και που ο εισηγητής παρουσίασε το άτομο δηλαδή που μίλησε πριν από μένα. Μιλάμε για το νέο κανονισμό της Europol ε, που υπέβαλε η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εγώ στην Επιτροπή μου πρόσφατα ε, σύστησα στην κυβέρνησή μου να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για αυτόν τον κανονισμό μέσα στην τρίμηνη περίοδο που είχαν υπό τις αλλαγές που εισήχθησαν στη συνθήκη της Λισαβόνας και που τους έδινε τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν ή όχι και καλωσορίζουμε όλος ιδιαίτερος στα πλαίσια των διαρκών εξελίξεων της Europol την απόφαση που ελήφθη νωρίτερα να δημιουργηθεί μέσα στη Europol ένα κέντρο για το κυβερνοέγκλημα. Δεδομένου, δεδομένης της ανάπτυξης του κυβερνοεγκλήματος και της σημασίας ε, για την οικονομία μας. Και πιστεύουμε ότι ήταν σημαντικό να βρίσκεται αυτό το κέντρο στο εσωτερικό της Europol. Επίσης, οι διοκτικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες με την Europol από ό,τι έκαναν στο παρελθόν και να χρησιμοποιούν περισσότερο και νωρίτερα τις, τους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας. Φυσικά, θα υπάρξουν ευαισθησίες για τον επιμερισμό τέτοιων πληροφοριών, το περιμένουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να το λάβουμε αυτό υπόψη στις διαπραγματεύσεις του νέου κειμένου του κανονισμού. Αλλά πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας αυτές οι ευαισθησίες να ξεπεραστούν και δίνουμε στην Europol και πρέπει να δίνουμε στην Europol ε, πιο διαρκείς και συνεχείς πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τους εγκληματίες. Ένα τμήμα της πρότασης Κομισιόν που μας απασχόλησε και μας ανησύχησε ήταν η ιδέα, στην οποία αναφέρθηκε και ο εισηγητής, της συγχώνευσης της Europol με τη C-Pol. Καταλαβαίνουμε γενικά ότι καλό είναι να συγχωνεύονται οργανισμοί και υπηρεσίε για να εξοικονομούμε χρήματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πειθόμαθα από τα επιχειρήματα σε αυτή την περίπτωση για αυτή τη συγχώνευση. Αυτέ τι αμφιβολίε τι έχουν και η πλειοψηφία των κρατών μελών όταν έγινε η πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδε. Και από ό,τι προέκυψε σαφώ και από την εισαγωγική παρουσίαση του εισηγητή, οι ανησυχίε αυτέ ε, βρίσκονται και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συγχώνευση δεν θα προχωρήσει. Γιατί οι Υπουργοί έδωσαν οδηγίε στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τι διαπραγματεύσεις αλλά χωρίς την ιδέα αυτή τη συγχώνευσης. Μας αρέσει όμως το τμήμα της πρότασης της Κομισιόν που ασχολείται με την κοινοβουλευτική εποπτεία της Europol και στην οποία αναφέρθηκε διαμακρόν ο εισηγητής. Είναι σαφές ότι στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της ποινική δικαιοσύνης οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπερδεύονται με, κάποιες, με πολλές από τις εθνικές αρμοδιότητες και επομένως θα πρέπει να βρούμε το σωστό μείγμα ε, κοινοβουλευτικής εποπτείας από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό το κείμενο της Κομισιόν. Και κατά την άποψή μου είναι καλό που επέλεξε ε, μία ελαφρά θεσμική δομή με συναντήσεις που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτή που έχουμε σήμερα α, ως μπούσουλα παρά να δημιουργεί νέες ε, και επαχθείς δομές. Ελπίζω να μην αποκλίνουμε από αυτό και θα πρέπει αυτή η κοινοβουλευτική εποπτεία να μην ελέγχει τις επιχειρησιακές πτυχές του έργου της Europol. Καμία από τις κυβερνήσεις μας και τα κοινοβούλια μας δεν θα δεχτούν ποτέ σε εθνικό επίπεδο αυτό, δεν θα δεχόταν αυτό σε εθνικό επίπεδο και άρα δεν πρέπει να το κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα κάτι εντελώ βρετανικό. Υπό τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η βρετανική κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κάνει opt-out από την νομοθεσία για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις που υπήρχε πρόλη αγώνας. Ε, δεν θα δεχτούμε επομένως τις αρμοδιότητες ε, από το 2014 και μετά της Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα. Εμείς ακούσαμε ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, ε, επαγγελματίες του κλάδου και η έκθεση, φτιάξαμε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση ε, δεν ε, έχει πιστικά επιχειρήματα για να χρησιμοποιήσει το opt-out. Ε. δεν φτάσαμε εύκολα σε αυτό το συμπέρασμα και έγινε ψηφοφορία. Θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία πριν από οποιαδήποτε απόφαση και στις τα δύο σώματα της Βουλής. Θεωρούμε ότι η Europol το, το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι πολύτιμο εργαλείο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, και η Βρετανία θα πρέπει να του γυρίσει την πλάτη και επομένως θα πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε η Βρετανία να παραμείνει εγγενές τμήμα της, ε, του μηχανισμού αυτού. Ευχαριστούμε, Λόρδε. Σας ευχαριστούμε για τον ε, τολμηρό τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τα επιχείρηματά σας. Μην ξεχνάμε τη μοναδικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις σχέσεις του, της χώρας αυτής με την συνθήκη της Λισαβόνας ε, στους χώρους της ε, δικαιοσύνης. Ξέρουμε το opt-in και opt-out της ε, Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας. Αποφασίστηκε ως ε, έσχατη καταφυγή για να μπορέσει η Λισαβόνα να τεθεί σε ισχύ τελικά και να μην υπάρξει μπλοκάρισμα. Κάνετε τις δηλώσεις σας, ε, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα εργαλεία συνεργασίας. Transporter. Για τα θέματα του σοβαρού διοσυνοριακού εγκλήματος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Περνάμε στην τρίτη παρέμβαση το βήμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Χάστινγκς, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση, θα σας εξηγήσω τους κανόνες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να συνεχίσω τις ε, συζητήσεις με την Επιτροπή σας και επίσης ε, χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να συναντήσω τα μέλη της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής. Για την ε, Europol τώρα θα ήθελα πρώτα να αναφέρω πως ε, ε, η επιχειρησιακή δουλειά της αστυνομίας γίνεται στο επίπεδο του κράτους μέλους. Αυτό είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή όμως. Οι επιχειρήσεις πλέον, οι αστυνομικές, είναι όλο και πιο πολύ διασυνοριακές και άρα αυτό σημαίνει όλο και μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, επιχειρησιακών και στρατηγικών και μεγαλύτερη ανάγκη τέτοιων ανταλλαγών πληροφοριών. Και εδώ πέρα ακριβώς υπησέρχεται η Europol. Η Europol παίζει ένα ρόλο υποστηρικτικό όσον αφορά την ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών για να διευκολύνει τις διοκτικές αρχές στο εθνικό επίπεδο. Η πρόταση της Κομισιόν της 1ης ε, Απριλίου έχει στόχο να ενισχύσει τον ρόλο και τη λειτουργία της Ευρωπόλ και άρα εισάγει κάποιες διατάξεις ενίσχυσης της προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων. Στην δική μας την ε, γνωμοδότηση που δημοσιεύτηκε τον Μάιο είπαμε πως ε, η στιβαρή προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, θα βοηθήσει στην διαρρεύνηση σοβαρών εγκλημάτων. Και είπαμε βέβαια πως χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη διερεύνηση κατάστασης στις δε σελίδες 34-38 της έκθεσης είχαμε αρκετές προτάσεις και χαίρομαι για το ότι ο εισηγητής ο κ. Διάρας Δεμέρα τις βρήκε χρήσιμες όπως είπε. Προσφάτως ε, υποβλήθηκε άλλη μία γνωμοδότηση από το κοινό εποπτικό φορέα της Ευρωπόλ που είχε συσταθεί στη δεκαετία του 90 με βάση μία σύμβαση ως το, το διακυβερνητικό ισοδύναμο της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Πρόκειται δηλαδή για εκπροσώπους των Εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν διαβάσετε τη γνωμοδότηση αυτή, μπορεί κάποιος να έχει την εντύπωση πως ε, διαφωνούμε στην αξιολόγηση της πρότασης. Και κάπου αυτό ισχύει, αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Η Europol τώρα έχει ένα στιβαρό καθεστώς προστασίας δεδομένων και θεωρούμε πως το επίπεδο αυτό δεν πρέπει να μειωθεί κάτω δένα τρόπο. Επίσης συμφωνούμε και στις δύο γνωμοδοτήσεις πως χρειάζεται κάποια βελτίωση. Μάλιστα, αν ε, τα δει κανείς προσεκτικά, θα δει πως ε, υπάρχουν πολλές παρόμοιες προτάσεις, καθώς ε, πως αυξάνονται οι ε, ικανότητες δεν χρειάζεται να μειωθούν οι δικλείδες ασφαλείας και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να ενισχυθούν. Ένας από τους τομείς που πρέπει να ενισχυθούν είναι η αρχιτεκτονική των πληροφοριών, όπου υπάρχει μια κάποια μεγαλύτερη ευελιξία η οποία χρειάζεται, αλλά δεν τονίζεται στην πρόταση η ανάγκη να συνεχίσουμε να καθορίζουμε τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών των αστυνομικών δεδομένων. Οπότε η αρχή του περιορισμού σύμφωνα με τον σκοπό είναι σημαντική και αυτό τονίζεται επίσης και στην ε, καθημερινή πρακτική της ε, Europol. Οπότε έχουμε κάποιες ιδέες για το πώς θα γίνει αυτό και πώς θα έχουμε περισσότερη ευελιξία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ανάγκη για μια αξιολόγηση αντικτύπου εκ των προτέρων πριν δημιουργηθούν νέα συστήματα πληροφοριών. Πρέπει δηλαδή να αξιολογηθεί αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και περιθώριο συζήτησης με, τις, ε, με τον επόπτη. Μιλώντας λοιπόν για υποπτία χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση η οποία επίσης απαιτεί και την εμπλοκή των εθνικών εποπτών δεδομένων από τη δική τους τη σκοπιά και υπάρχει στενή αλληλεπίδραση. Και τέλος νομίζω πως ε, συμφωνούμε και στο ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί η πρόταση με το νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων που είναι μια άλλη παράλληλη σοβαρή δραστηριότητα και περιλαμβάνει μια οδηγία και έναν κανονισμό με κάποιες καινοτόμες ιδέες που πρέπει βεβαίως να ενταχθούν κάποτε στους κανόνες της Ευρωπόλ. Πού διαφέρουμε τώρα, και εδώ πέρα θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα, ότι δηλαδή στο πλαίσιο της ανάγκης για μια πιο ενισχυμένη υποπτική δομή. Έχει περάσει η στιγμή να περάσουμε από την διακυβερνητική προσέγγιση της δεκαετίας του 90 στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την έννοια της εποπτείας ε, από την δική μου υπηρεσία. Εμείς εποπτεύουμε 50 ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς. Έχουμε τις αρμοδιότητες από τον νόμο και έχουμε όμως ελάχιστους πόρους, ε, περιορισμένη ανεξαρτησία, οπότε καλωσορίζω την πρόταση να υπάρξει ισχυρή εποπτεία. Αλλά τονίζω αυτό μπορεί να λειτουργεί στην πράξη μόνο αν υπάρχει στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και όπως ερμηνεύω εγώ την πρόταση αυτό υπάρχει οπότε θα πρότεινα να διατηρήσουμε αυτή την αλλά να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ένα πρακτικό παράδειγμα. Ροή δεδομένων ε, στην ε, Europol. Πάνε τα δεδομένα από τη Europol στα κράτη-μέλη. Η Europol συλλέγει πληροφορίες και από άλλες πηγές και από ιδιωτικές πηγές κάποια στιγμή και καθώς το βλέπουμε συνολικά το ζήτημα θα πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να ξέρουμε και ολόκληρο τον αντίκτυπο. Εάν, εάν χρειαστεί κάτι, εάν πάει κάτι στα, εθνικά, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, εάν αφορά τα εθνικά δικαστήρια είναι εθνική υπόθεση. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκς. Είπαμε, συζητούμε τις προκλήσεις ε, της Europol και πιο συγκεκριμένα τις προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, λάβοντας μπορείς το άρθρο 88 για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και ένα τέταρτο μέλο του πάνελ που θα έρθει να μα κάνει μια παρουσίαση όπω είπαμε και θα το δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο, γιατί καθυστέρησε λόγω της κίνησης. Είναι ο κύριος ε, Ντίτιχ Νόημα, τελικά καταφέρατε να έρθετε και καλώς ορίσατε. Αν θέλετε μπορείτε να κλείσετε αυτό το, το γύρο παρουσιάσεων και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. He is head of the Business Corporate Division in Europol. He's representing thus the agency. Εκπροσωπεί την Europol ο κύριος Νόημαν. Thank you, Mr. Chairman. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί κύριοι ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές, πρώτα πρώτα να ζητάω συγγνώμη, διότι καθυστέρησα να φτάσω. Τέλος όταν έφτασα ακριβώς την ώρα που ήταν να μου δώσετε το λόγο. Ε, αυτό κάνει και η αστυνομία, έρχεται ακριβώς τότε που χρειάζεται. Να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους της τροχίας των Βρυξελών για να ρυθμίσουν όλα αυτά τα μποτιλιαρίσματα. Πάντως ευχαριστώ που με καλέσατε γιατί θεωρώ τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Ο διευθυντής μας δεν μπόρεσε να έρθει και έτσι ε, αυτού σας μιλώ εγώ σήμερα όσον αφορά α, αυτή το νέο νομοθέτημα, τη νέα νομική βάση. Πάντοτε είναι σημαντικές συναντήσεις αντισημερινή. Θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπή θέλει να κάνει πιο αποτελεσματική τη Europol με αυτό το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Δεύτερον, αυτό το σχέδιο κανονισμό περιέχει πολλές καινοτομίες, ε, καινούργια διάρθρωση. Εγώ ως νομικός θεωρώ ότι είναι πιο εύχριστο, έχει περισσότερη διαφάνεια και κατά τρίτον τώρα το καινούριο πλαίσιο να μας κάνει πιο αποτελεσματικούς. Και επίσης για την καταπολέμηση σοβαρού κλίματος και τρομοκρατία μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τα κράτη-μέλη. Ο κανονισμός επιφέρει κάποιες θετικές αλλαγές. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υπάρχει πιο πολύ επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα καλύτερη, ευκολότερη τέλο πάντων συμμετοχή σε κοινέ έρευνε από πλευρά Europol, καλύτερη επικοινωνία με τι ε, συναρμόδιε αρχέ, καλύτερη ροή πληροφοριών. Άμεση διεύρυνση πληροφοριών από τα κράτη-μέλη προ την Europol και επίση ευκολότερη χρηματοδότηση στη δραστηριοτήτων από πλευρά κρατών μελών ή από πλευρά προπολογισμού τη Europol. Μια από τι βασικές καινοτομίε του καινούργιου νομοθετήματο είναι αυτό που ονομάζουμε ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων. Και έτσι τώρα θα ανανεώσουμε τον δοκιμασμένο μεν μηχανισμό, ο οποίος όμως έχει ηλικία 15 χρόνια. Γιατί πρέπει τώρα είναι άλλα τα, αυτά που απαιτεί η σημερινή καταπολέμηση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Οι σημερινές απειλές επομένω έχουν πιο δυναμικό χαρακτήρα, πιο διεθνή χαρακτήρα. Οι προηγούμενες δεκαετίες είχαμε μεγαλύτερη κατάτμιση το, της διαχείρισης των δεδομένων. Όταν η Europol είχε πολύ συγκεκριμένε απειλές να αντιμετωπίσει όπως ας πούμε λαθρεμπόριο κοκαίνης ή ε, η διακίνηση παράνομη ανθρώπων ήταν διαφορετικά. Τώρα έχουμε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες και επομένως είναι, έχει πιο πολλαπλό χαρακτήρα η εγκληματική δραστηριότητα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε τις πληρω... τους περιορισμούς που μας παρουσιάζει η σημερινή ρυθμίση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα επιμέρους ε, συστήματα πληροφοριών, θα πρέπει να μην εμποδίζονται οι αναλυτές μας να κάνουν όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ των δεδομένων που με σύνομο τρόπο ε, συλλέγονται από την Europol. Οπότε γι' αυτό και η εντύπωσή μας είναι, αλλά και η εμπειρία μας είναι, ότι μέχρι τώρα είχαμε φραγμό στο να μπορέσουμε να αποδώσουμε όσο γίνεται καλύτερα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Άρα, τώρα έχουμε κάποιο λογικό διαχωρισμό του εδώ λίγο με τον, με τον σκόπο της δουλειάς μας κάθε φορά, αλλά θα έχουμε και, όλα, και όλες τις, ε, τις, τις για την σωστή διαχείριση. Τα κράτη-μέλη συνεχίζουν βέβαια να έχουν ε, την κυριότητα αλλά και έλεγχο στα δεδομένα τους. Θέλουμε το ύψιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Άλλωστε, θεωρούμεθα ότι από όλες τις ευρωπαϊκές αστυνομίες εμείς έχουμε την καλύτερη προστασία δεδομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα ανάλογα, ε, ανεξάρτητα μάλλον από την ε, δομή λειτουργία τη διαχείριση, θα διέπονται από αυτή την αρχή της ε, προστασίας των δεδομένων, οπότε δεν πρόκειται να πέσει το επίπεδο προστασίας, μάλλον θα βελτιωθεί. Άλλωστε, τώρα θα έχουμε απλούστευση τη της επεξεργασίας, απλούστευση των συστημάτων, μόνο μια φορά αποθήκευση διάσωση των δεδομένων και θα έχουμε τους ελέγχους και ό,τι προβλέπεται για την προστασία αυτών των δεδομένων. Έχουμε την οδηγία 44 για την προστασία των δεδομένων. Και αυτή λαμβάνεται υπόψη και όπως είπαμε επί 15 έτη η προστασία λειτουργήσε μια χαρά. Η ε, οι αρχές που διαπνέουν την βέβαια δεν φτιάχτηκαν για σκοπούς ιδιωτικής αρχής. Άρα θα πρέπει να γίνει προσαρμογή. Για να δούμε πώς θα υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα. που μας αφού θεωρούμε ότι είναι αρκετά ε, υψηλό το επίπεδο προστασία και ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, ίσως ε, αλλαγές εκβάθρων δεν χρειάζονται. Πάντως, όσον αφορά τον νέο οργανισμό, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την προτινόμενη συγχώνευση με την ΣΥΠΟΛ. Δεν μπορώ να πω πολλά, καταλαβαίνετε γιατί. Τα κράτη-μέλη έχουν την άποψή τους και το Ε, μελετούμε τις προτάσεις, δεν μπορώ να πω άλλα, σχόλια, πάντως οπότε χρειαστεί ενημέρωση για να γίνει οριστική διαμόρφωση της πρότασης, εμείς να συνεργαστούμε. ευχαρίστως Οι προτάσεις για υποχρεώσει λογοδοσία, αλλά και για περισσότερη διαφάνεια μα βρίσκουν σύμφωνο. Θέλουμε να υπάρχει τακτή ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα με το, Εθνικό, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ συχνά άλλωστε ερχόμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολύ στενή και επικοδομητική σχέση με το Κοινοβούλιο. Για ακριβώ όπω ε, και σήμερα θεωρούμε ότι αυτά είναι μια ευκαιρία να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για το έργο μας. Εάν έχετε πιστεί ότι το έργο τη Europol ε, είναι χρήσιμο, τότε μπορείτε να μας ε, βοηθήσετε και στη συνεργασία με τους εθνικούς βουλευτές και ε, προβάλλοντας το έργο μας στους ψηφοφόρους σας, στους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε, θεωρούμε θετικό το σχέδιο αυτοκανονισμού που όταν εγκριθεί θα έχουμε μια νομική βάση ώστε να έχουμε αναβαθμισμένη συνεργασία. Και έτσι μπορούμε να ενημερώσουμε Εθνικά Κοινοβούλια, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις λεπτομέρειες του έργου μας, ας πούμε, ε, αναλύσεις κινδύνου, στατικές αναλύσεις, εκθέσεις γενικής κατάστασης, μελέτες, ακόμα και τις ε, ρυθμίσεις και τις συμφωνίες που κάνουμε με τους ε, συνεργάτες μας, τους τρίτους. Βεβαίω και το έχουμε και το πρόγραμμα εργασία, να δούμε πώ θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίση θα εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ε, στον διορισμό των στελεχών, εκτελεστικών διευθυντών κλπ. Και επίση θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το ότι αυτό ο κανονισμό ε, προβλέπει τη δυνατότητα να λάβει επίσημο χαρακτήρα η προσβασιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε, σε, σε, σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπάρχουν ε, και αυτό θα ολοκληρωθεί μόλις προβούμε στις τελικές ρυθμίσεις συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, η σύντομη εισηγησή μου εδώ ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονικό όριο το οποίο έχετε θέσει και ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. ακούσαμε κάποια στοιχεία. Τώρα, με βάση τους κανόνες αυτής της συζήτησης θα δώσουμε το λόγο σε μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων ανά ομάδες δύο ή τριών και συνεχεία σε έναν Ευρωβουλευτή, ούτως ώστε να ακούσουμε από διαφορετικά άτομα τις απόψεις τους για τον προτινόμενο κανονισμό. Για την αστυνομική συνεργασία και επίσης την εμπλοκή ε, των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επίσης, θα δώσουμε, τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ματάη από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Κυρία ή κύριος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο της Ευρώπης δέχτηκε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Τώρα έχει περάσει ε, ένα κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ε, Στοκχόλμη. Χρειαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα και καθοδήγηση από το Συμβούλιο. Για την Ουγγαρία η λαθρομετανάστευση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα για να την καταπολεμήσουμε. Γιατί η λαθρομετανάστευση από τον Νότο και τα Ανατολικά διοχετεύεται μέσω της Ουγγαρίας στην περιοχή του Σέγγεν. Υπήρξε ε, σημαντική αύξηση από το 2008 αυτού του τύπου της ε, το 2010 και το 2011 είχαμε αύξηση 30 με 40% της ε, παράνομης μετανάστευσης. Και ακόμα πιο εντυπωσιακή ε, αύξηση που έφτανε στο 150% πρόσφατα. Υπήρξαν όμως και κάποιες θετικές εξελίξεις. Η Frontex και η Κομισιόν μας ανακοίνωσαν τις θετικές εξελίξεις αλλά έχουμε την αίσθηση ότι στην Ουγγαρία ε, πέφτουμε θύματα της λεγόμενης δευτερογενούς μετανάστευσης. Το πρώτο τρίμηνο είχαμε 658% αύξηση σε αιτήσει που υποβάλλονταν για το καθεστώς του πρόσφυγα. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ε, καταχρήσεις του συστήματος. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ εντατικά μαζί με τα κράτη-μέλη και τις ε, τρίτες χώρες που συναποτελούν το πρόβλημα. Στην έκθεση του 2012 της Frontex για τα εξωτερικά χερσαία σύνορα η Ουγγαρία είχε το δεύτερο υψηλότερο αριθμό μεταναστών Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την Αυστρία και τη Σερβία και επεκτείνουμε όλο ένα αυτή τη συνεργασία με κράτη-μέλη και τρίτες χώρες από τα οποία προέρχεται, τρίτα κράτη από τα οποία προέρχεται η λαθομετανάστευση. Πρέπει λοιπόν, επειδή ακριβώς αυτό το πρόβλημα δεν δημιουργείται σε ένα κράτος, όλοι μαζί να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για να το αντιμετωπίσουμε. Η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθάει την Ουγγαρία για να παίξει το ρόλο του φύλακα αγγέλου σε αυτές τις δραστηριότητες, σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε γραφεία, έχουμε εστιακά σημεία, έχουμε αποσπασμένους υπαλλήλου από άλλες χώρες για να συνεργαστούμε μέσω αυτών με αυτές τις χώρες και η Ουγγαρία κάνει πολλά για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των ροών λαθρομετανάστευσης και βεβαίως να βοηθήσει για την σύλληψη των εγκληματιών που υποθάλπουν αυτή τη μετανάστευση. Τώρα, θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους που θέλουν να πάρουν το λόγο, αλλά η κυρία Λεμπάγη ε, θα έρθει εδώ στις 10.40 που είναι Γενική Διεύθυνση από τη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης και την, επίτροπο, ε, την αρμόδια επίτροπο Σεσίλια Μάλστρομ. Επομένως όλοι μας ας αυτοσυγκρατηθούμε λίγο στις ομιλίες μας, δύο-τρία λεφτά θα έλεγα ο καθένας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πρώτο γύρο και δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το σφυράκι. Η κυρία Κρέγκερ από το Κροατικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Είσαστε, είσαστε κύριος. Ναι, ναι, κύριος. Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Ο κύριος Κρέγκερ, λοιπόν. Και u Europsku uniju. Κυρίες και κύριοι. Η Κροατία θα ενταχθεί πολύ σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές τις μέρες η Κροατία υιοθετεί νόμους οι οποίοι αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις. Και είμαστε σε φάση προσαρμογής της νομοθεσίας μας με βάση τα όσα δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία είναι πολύ ανήσυχη και συμμεριζόμαστε και κατανοούμε απόλυτα όλα τα προβλήματα που έχουν οι όμορες χώρες για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Επομένως, η συνεργασία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ζητούμε ένα υψηλότερο βαθμό συνεργασίας με όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμούμε να επιτύχουμε ένα βαθμό συνεργασίας που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα αυτό για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Φερρυπίν κατάσχεση, η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί με εγκληματική δραστηριότητα και η οριστική τους δίμευση και άλλες μορφές ε, συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Από την εμπειρία που έχουμε μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι με πολλές χώρες είχαμε πολύ καλή συνεργασία σε διμερές όμως επίπεδο. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες που μας επέτρεψαν αυτή την ε, συνεργασία με αστυνομικές αρχές διαφόρων χωρών. Έχουμε θαυμάσια εμπειρία σε ό,τι αφορά τις δράσεις, ε, σε ό,τι αφορά την ε, δραστηριότητα διαφόρων αστυνομικών αρχών, γειτονικών ή άλλων χωρών, που συνεργάζονται με, τις, με την κροατική αστυνομία. Ήταν πολύ καλή αυτή η συνεργασία. Ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι πιο έντονη για να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Ελπίζω ότι με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια που παραμένουν ακόμα. Δεν θέλουμε να διευκολύνουμε το βίο των εγκληματιών. Επειδή μπορούν να περνάνε τα σύνορα εύκολα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος ελεύθερος, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει τις χέρειες για το έργο των αστυνομικών αρχών. Ο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Κύριε σας ευχαριστώ. Είμαι εκπρόσωπος των συντηρητικών του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτό το θέμα. Να σας πω το πόσο καλωσορίζουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά είναι χαρακτηριστική νομίζω του πώς συζητάμε με ανοιχτό τρόπο τις επιχειρήσεις της Europol, την οποία εκτιμούμε όλοι πάρα πολύ, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ως ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις ε, έρευνες ε, ε, ζητήματα εργονομένου εγκλήματο. Και θα ήθελα επίση να συγχαρώ τον Λόρδο Χάνη για αυτό το οποίο γίνεται στην Βουλή των Λόρδων, όπου εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά όλα τα ζητήματα, ειδικά τον νέο κανονισμό και δίνουν πάρα πολύ καλές συμβουλές στην Βρετανική κυβέρνηση. Και νομίζω πως ε, το θέμα ενδιαφέρει και άλλες χώρες και φαίνεται και από την προσέλευση σήμερα Δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα αφορά το θέμα της εποπτείας και το άλλο τα προσωπικά δεδομένα. Για την εποπτεία. Προφανώς αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στην συνθήκη το άρθρο 88 το οποίο ορίζει την επιχειρησιακή δράση της Europol, η οποία πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των αρχών των κρατών μελών ε, ε, στην επικράτεια των οποίων γίνονται οι έρευνες και των ε, αρμοδίων αρχών. Και παρά το ότι σέβομαι ιδιαίτερα το έργο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τη νέα κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν εάν περάσουν αυτά τα θέματα, μου φαίνεται πως δεν θα έπρεπε να είναι αποκλειστικές αυτές οι αρμοδιότητες και να μην έχουμε την διαφάνεια που είχαμε μέχρι τώρα. Ε, υπάρχει κάποια δυσκολία γιατί ε, βεβαίως σας γνωρίζουμε ε, είστε τακτικός ε, προσκεκλημένος εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο, οπότε εσείς επιδεικνύετε διαφάνεια, αλλά δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Πρέπει να έχουμε σωστή ισορροπία και στο μέλλον όσον αφορά αυτές τις αρμοδιότητες. Για τα δεδομένα τώρα. Να πω πως με τις ανησυχίες που είχαμε μετά τη συζήτηση για το πρίσμα στις ε, ΙΠΑ, το οποίο το συζητάμε ε, όλη τη βδομάδα που μας πέρασε και θα μας απασχολήσει για καιρό ακόμα, νομίζω πως ανησυχούμε και με τον νέο κανονισμό και οδηγία προσωπικών δεδομένων, ανησυχούμε για τα δεδομένα που συλλέγονται για τους πολίτες της Ευρώπης και η χρήση των δεδομένων αυτών θα πρέπει να προστατεύεται. Βεβαίως υπάρχει ο υπόπτης προστασίας δεδομένων, αλλά ειλικρινά νομίζω πως υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η διοκτικές ε, αρχές θα πρέπει να μπορούν βεβαίως να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτό το οποίο δεν θέλω να δω είναι να έχουμε τέτοιους κανονισμούς που να αποτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ αστυνομιών και λοιπόν διοκτικών αρχών. Γιατί ξέρετε, τα δεδομένα στον εμπορικό κόσμο ε, διακινούνται πολύ πιο ελεύθερα από ότι ε, τα δεδομένα που θέλουμε εμείς για ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας. Πρέπει λοιπόν να το προσέχουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι διακεκριμένο το πάνελ μας, μας καθησυχάζουν και εγώ και οι συνάδελφοί μου οπωσδήποτε θα στηρίξουμε την Europol και το μάλλον της και την εμπλοκή των κρατών μελών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρω πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια και εντός της ε, Ευρωπόλ, αλλά βεβαίως υπάρχουν και ανησυχίες που έχουμε όσον αφορά την χρήση ε, των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των πολιτών μας. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτά υπόψη και γι' αυτό ε, είναι καλοδεχούμενη και η σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Περνάμε ξανά στους εθνικούς βουλευτές. Έχουμε κάποιους Ιταλούς βουλευτές. Κρίνη πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Ε, είμαστε δικοί στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εγκληματικότητας. Συμφωνούμε και με το πάρτιμα 1 του σχεδίου κανονισμού. Όμως θα πρέπει να οριοθετήσουμε τα όρια της συνεργασίας. Δεν θα πρέπει να έχουμε αλληλεπικαλύψεις με άλλα κανάλια συνεργασίας που υπάρχουν ήδη. Και να αποφύγουμε η Europol να γίνει ένας ε, υπερκρατικός ε, οργανισμός. Να παραμείνει στο πλαίσιο που πρέπει. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Europol από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και όχι μόνο να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης, να έχετε εσείς την δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες του αργού της Europol. Θα πρέπει να γίνεται και μεγαλύτερος άμεσος έλεγχος από τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει ο έλεγχος να περιορίζεται μόνο στην πρόσβαση των δεδομένων που έχει η Europol. Επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ε, μοιραζόμαστε ε, δεδομένα με ιδιωτικούς φορείς όπως προβλέπει ο κανονισμός. Όλα αυτά θα πρέπει να προσδιοριστούν πολύ πιο ενδελεχώ. Επίσης, όπως υπόθηκε, είναι σημαντικό η Europol μεταξύ των στόχων της να έχει το στόχο την πρόθεση τα δεδομένα που, έχουν, που έχουν τα κράτη-μέλη να είναι μεταξύ τους ώστε να τον πιο συμβατά για να υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερου διαλόγου και ομοιογένειας των δεδομένων και για να μπορούν τα δεδομένα αυτά να αξιοποιούνται από το ένα κράτος από τα διάφορα κράτη, με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Επίσης πρέπει να περάσουμε από μια κουλτούρα όπου όλες οι πληροφορίες βρίσκονται σε υπόθεμα χάρτου, σε μια κουλτούρα ε, ηλεκτρονικού υποθέματος. Επίσης. Και βάσεων δεδομένων βέβαια. Πρέπει να δημιουργούμε βάσεις δεδομένων. Επίσης, ε, τα όσα είπε ο Βρετανός συνάδελφος από την ε, Βουλή των Λόρδων είναι πάρα πολύ θετικά. Θεωρούμε ότι είναι θετικό. Ε, και εδώ μιλάω εξ ονόματος του, του κινήματος Cinque Stelle, πέντε αστέρια. να δίνονται εξηγήσει, συμφωνώ με, το, με αυτό που λέει ο κανονισμό, να δίνονται εξηγήσει σε περίπτωση που δεν ξεκινάνε ή δεν προχωρούν διάφορε έρευνε. Πρέπει να ξέρουμε γιατί. Επίσης, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα λόγω του καονισμού ε, στην αυτονομία ε, των δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Για τη συγχώνευση του ΣΕΠΟΛ και της Europol, αντίθετα από ό,τι είπαν οι προλαλήσαντες, εμείς είμαστε θετικοί. Θέλουμε να συγχωνευτούν τα δύο αυτά όργανα, ΣΕΠΟΛ και Europol. Ε, αυτό βέβαια είναι η άποψη του κινήματος που εκπροσωπώ, ο κύριος Φαμιλιέτη. Καλημέρα. Έχουμε μια πολύτιμη ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε απόψεις για ένα θέμα ε, μεγάλης πολιτικής σημασίας, ε, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της Europol. Νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση πηγαίνει προς την πολιτική ένωση των ευρωπαϊκών χωρών. Η, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του, της Ιταλικής Βουλής εξετάζει τον εν λόγω καονισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας δοθούν όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να τον εξετάσουμε. Η Europol μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε σημαντική πρόοδο, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας. Και σε επίπεδο ερευνών και σε επίπεδο ε, επιμερισμού των δεδομένων. Ε, υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων ε, με σκοπό να προστατεύσουμε φυσικά τα εν λόγω άτομα. Το διασυνοριακό έγκλημα είναι το πιο σοβαρό, το πιο επικίνδυνο έγκλημα και νομίζω ότι εκεί μπορεί να βοηθήσει η Europol να, με τον επιμερισμό και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια, κάποιοι προβληματισμοί, ε, κυρίως στους εξή Καταρχάς, δεν είναι σαφές αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει στη Europol πέρα από ρόλους συντονιστικούς και αρμοδιότητες επιχειρησιακές. Αν ναι, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον κίνδυνο αύξησης ε, του ρόλου της ε, Europol και αυτό μπορεί να δημιουργήσει συγχύσεις ή αμφισημίες. Δεύτερον, και εδώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον ε, Αγκουστίν Δίας Δεμέρα, μπορεί να είναι άστοχο να συγχωνεύσουμε τη ΣΕΠΟΛ με τη Europol και να την εντάξουμε στο εσωτερικό της Europol. Ε, ο στόχος βέβαια είναι να εξοικονομήσουμε χρήματα, αλλά μπορεί όμως ε, θυσιάζοντας τη ΣΕΠΟΛ η οποία μέχρι στιγμής λειτουργήσε πάρα πολύ και μας βοήθησε για να καταπολεμήσουμε διάφορες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, ίσως γι' αυτό λοιπόν να μην είναι σωστό να προβούμε σε αυτή τη συγχώνευση. Επίσης, η διαχείριση, η διακυβέρνηση, αν θέλετε, της Europol δεν είναι η βέλτιστη δυνατή. πολύ συχνά πολλαπλασιάζουμε οργανώσεις χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, ενώ σε αυτή την περίπτωση την Europol και σε ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να προβούμε σε αυτή τη συγχώνευση. Επίσης, ο δημοκρατικός έλεγχος της Europol. Η... Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος ο ρόλος της Europol, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα δεδομένα που επεξεργάζεται. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται η υπηρεσία αυτή για να, υπάρχουν, να μην υπάρχει περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων αυτών. Επομένως, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο εισηγητής Δίεστε Μέρα. Και συμφωνώ επίσης και με τα όσα είπε ο κύριος Χάστινγκς. Ε, ο κύριος Δίαντε Μέρα είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα διακοινοβουλευτική με σκοπό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και θα πρέπει να υπάρχει πραγματική, μια πραγματική εγγύηση ε, σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και να υπάρχει συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο η πρόταση καονισμού είναι ανεπαρκής. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας το άρθρο 88 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν σοβαρότατες αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Ο κ. Άλμπρεχτ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο επόμενος ομιλητής. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή απόψεων. Και ε, τώρα σε σχέση με τη Europol θεωρώ πως πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, να κάνει τη δουλειά της ε, και να ενισχύσουμε και την διασυνοριακή συνεργασία. Εμείς, ε, κατά την άποψή μου, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις κοινέ ομάδες έρευνας που πρέπει να ενισχυθούν για να υπάρξει η άμεση συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών της Ευρώπης και για να βελτιωθεί η δουλειά τους. Τώρα, όσον αφορά τον κανονισμό, πολλές από τις ε, προτάσεις ε, του κυρίου Δίας Δεμέρα ακούγονται πολύ σημαντικές, ειδικά το ζήτημα της ε, κοινοβουλευτικής εποπτείας είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο και στο πλαίσιο της σημερινής ε, συζήτησης νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα, οπότε υπάρχει νομίζω. Ε, πρέπει να υπάρχει κοινό έλεγχο από εθνικού ε, και ευρωπαίου βουλευτέ για το πώ δουλεύουν αυτοί οι φορεί, αλλά βέβαια και η εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί. Θεωρώ πως γίνεται τόσο αποδεκτή δουλειά της ε, Europol ακριβώς γιατί υπάρχουν και σοβαρές δικλίδες ασφαλείας, ειδικά για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλω να τονίσω αυτά τα οποία είπε ο Πίτερ Χέστινγκς πως ε, ναι. δεν πρέπει να μειωθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι γιατί μπορούμε νομίζω να δείξουμε κάποια εμπιστοσύνη και να πούμε πως η Europol αποτελεί και ένα παράδειγμα για τις εθνικές αρχές. Γιατί εάν θέλουμε πραγματικά να τονίσουμε τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αστυνομικών αρχών στα κράτη-μέλη πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη πως υπάρχει πραγματική και ίση προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικά στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, που είναι η καθημερινή δουλειά της έρευνας και των ομάδων έρευνας και πρέπει άρα να έχουμε κοινά πρότυπα και αυτό θέλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, ακριβώς εδώ πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις ε, δικές μας προδιαγραφέ με τις προδιαγραφές Ευρωπόλ με αυτές των κρατών μελών. Και θέλω να τονίσω άρα και τη νέα οδηγία ε, προσωπικών δεδομένων ε, στον τομέα της αστυνομία που δεν προωθείται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο και όπου ελπίζω πραγματικά οι συνάδελφοι των Εθνικών και του να ασκήσουν πίεση προς αυτή την ε, κατεύθυνση για να υπάρξουν αυτές οι ανταλλαγές. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, έγιναν κάποιες ερωτήσεις και σχόλια ε, όσον αφορά τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και ο κύριος Δίας Δεμέρα πρέπει να φύγει πριν από το τέλος του πρώτου γύρου, οπότε ας ε, του δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει και μετά τα επόμενα 20 λεπτά θα συνεχίσουμε με τους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Δίας Δεμέρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα. Στις 5 στην Ισπανία πρέπει να παρθώ σε μια εκδήλωση τρογγυλή τραπέζι, μια συζήτηση τέλο πάντων. Οπότε από τώρα σα ζητώ συγγνώμη που θα σκοτώ να φύγω. Ε, Πάντω πρέπει να ευχαριστήσω για όλε τι παρατηρήσει Όλα αυτά αποτελούν μια επικοινωνία. Είτε πρόκειτο για ε, παρατηρήσεις, είτε πρόκειτο για ερωτήματα και διαμορφώνονται δύο άξονες, δύο πλευρές, σύμφωνα και με τις δύο. Πρώτα-πρώτα έχουμε στον άξονα που αφορά την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά την ε, ασφάλεια, όσον αφορά τη λειτουργία μιας ιδιοκτική αρχής. Πρόκειται για την κλασική προβληματική δηλαδή. Το τι θα κατησχίσει. Η ελευθερία ή η ασφάλεια. Συχνά λέμε ότι προηγείται η ελευθερία ή οι ατομικές ελευθερίες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ασφάλεια εάν δεν διέπεται η εξασφάλιση της ασφάλειας, ας πούμε, από την, το σεβασμό της ελευθερίας. Και οριοθετεί όλες τις δραστηριότητες σε μια δημοκρατία το κοινοβούλιο. είπαμε ότι έχει ένα στεγανό σύστημα προστασία δεδομένων η Europol και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Χάστινγκς και με αυτά που είπε ο κύριος Άλμπεχτ ε, όσον αφορά την προστασία δεδομένων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί ο κύριος Άλμπεχτ μπορεί να είναι νέος, το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Και ο κύριος Χάστινγκς. Είπαμε όμως ότι έχουμε αυτή την ε, ομάδα του κοινοβουλτικού ελέγχου. Πώς θα συνεργάζεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόκειται για μέσο εξασφάλισης εγγύσεων και για την προσοχή των δεδομένων αλλά γενικότερα για τις δραστηριότητε που ρυθμίζει ο εν λόγω κανονισμός και θα τις ασκεί η Europol. Μπορεί να φαίνεται κάπως πρόημο, αλλά μπορείτε να δείτε τι θέλω να προτείνω, πώς θέλω να διαμορφώσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι το ίδιο πνεύμα που διαπνέει τις ε, συζητήσεις που κάνουμε πάντα για αυτά τα ζητήματα. Τα είπαμε και στην προηγούμενη θητεία και, τότε είχαμε κάνει επίσης ε, κάποιες συνεδριάσεις, κάποιες ακροάσεις που ήταν μονογραφικού χαρακτήρα, δηλαδή αφορούσαν ε, αποκλειστικά το γενοκτικό έλεγχο τη Europol. Επομένω με θεμέλιο, με αφετηρία αυτή τη συζήτηση θα προχωρήσουμε. Και φυσικά πρέπει να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ το έργο τη Europol. Και θέλω να πω, ιδίω στου ε, Βρετανού συναδέλφου ότι πριν διαμορφώσω την ε, πρότασή μου μίλησα με πάρα πολλού και ιδίω μίλησα με την Βρετανική κυβέρνηση. Και η Βρετανική κυβέρνηση επίσης εκτιμά το έργο της Europol. Φυσικά και πολλές άλλες κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση θέλουν να διατηρηθούν οι εθνικές αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ακριβώς όπως ξεκίνησε την εισήγησή του ο Πίτερ Χάστινγκς. Όμως θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση αυτών των εθνικών αρμοδιοτήτων με τις αρμοδιότητες της, ε, της Europol. Με γνώμονα την ασφάλεια και την ε, συνεργασία, την καλύτερη συνεργασία. Και πολύ σωστά τα είπε και ο Ιταλός συνάδελφος. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρηματικές αρμοδιότητες, αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτές οι αρμοδιότητες, θα ασκούνται από τις κοινέ ομάδες. Δεν θα έχει την ε, διοίκηση η Europol ποτέ. Θα είναι ε, συνδιοίκηση κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο θα ισχύει. Είμαστε στη διάθεσή σας, με email μπορούμε να βιονίσουμε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Οπωσδήποτε θα ήθελε να θα ήθελα να μιλήσουν και τα υπόλοιπα μέλη του πανέλα αλλά θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με τους βουλευτές και σας θυμίζω πως ε, σε 10 λεπτά θα έρθει η κυρία Λεμπάη και η κυρία Μαλευθρόμ. Οπότε παρακαλώ να περιοριστείτε στα 2 λεπτά. Το ρόλο έχει ο κύριος Γκρουλίχ από την Τσεχία για 2 λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την διακοινοβουλευτική αυτή συνεδρίαση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη κατά την απόψή μου. Έχω κάποια προσωπικά σχόλια. Και βεβαίω θα βαστώ στις θέσεις της τσεχικής ε, γερουσίας. Είναι σαφές ε, πως χρειαζόμαστε κάποιες κοινοβουλευτικέ διαδικασίες για την υποπτία της Ευρωπόλ και του έργου της. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τον κανονισμό, αλλά το μέλλον της Ευρωπόλ και του ΣΕΠΟΛ είναι κάτι ε, για το οποίο έχουμε τις αμφιβολίες μας. Γι' αυτό υπάρχει και κριτική από τα κράτη-μέλη και από την Τσεχία. Γι' αυτό νομίζω πως είναι καλή ιδέα να ξαναδούμε νομίζω την αρχή ιδέα και να την επανυποβάλλουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπαριθμών 1. Δεν είναι σωστό σε ένα τέτοιο έγγραφο να γίνονται αλλαγές μόνο μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και να σχολιάζουν τα κοινοβούλια μια παλαιότερη έκδοση. Σας ευχαριστώ κύριος Βλαχογιάννης από την Ελλάδα. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, προσεγγίζουμε θετικά το θέμα του νέου κανονισμού και πραγματικά έχει παραχθεί ένα σημαντικό έργο για το οποίο πρέπει να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που πάντα πρέπει να ασκείται και πάντα πρέπει να λογοδοτούν όλες οι αρχές στους εκπροσώπους του λαού. Είμαστε υπέρ των κοινών επιχειρήσεων. Το διασυνοριακό έγκλημα ξέρουμε ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και μάλιστα προηγείται τεχνολογικά της τεχνολογίας γενικότερα των κρατών μελών και η συνεργασία είναι άκρος απαραίτητη. Θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο από την Ουγγαρία για το μεγάλο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Η χώρα μας, ξέρετε, δέχεται το 70% του όγκου των λαθρομεταναστών από Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή. Και φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κατά groups δεν έρχονται στην τύχη. Κάποιοι τους διακινούν Κάποιοι τους καθοδηγούν και κάποιοι τους εκμεταλλεύονται. Άρα ένα έγκλημα σύγχρονου δουλεμπορίου πρέπει να παταχθεί και δεν μπορεί να παταχθεί μόνο από ένα κράτος. Απαιτείται κοινή συνεργασία και κοινέ επιχειρήσεις γιατί αυτοί, ας μην γελιόμαστε, δεν έχουν προορισμό μόνο ένα κράτος μέλος. Αυτοί έρχονται για μια καλύτερη πατρίδα και θα τη βρουν προφανώς, πιστεύουν, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο σε ένα κράτος μέλος. Διατηρούμε επιφυλάξει ε, σε ό,τι αφορά την ε, συνένωση των δύο οργανισμών, της Europol και της ΕΠΟΛ. Και μάλιστα έχουμε εκφράσει και την βούλησή μας σε περίπτωση που η ΣΕΠΟΛ με την κατασταθεί να τη φιλοξενήσουμε γιατί έχουμε εγκαταστάσεις και θα μπορούσαμε πραγματικά να συνεισφέρουμε κι εμείς σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μορένο από την Ισπανία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συνεργασία των διοικητικών αρχών στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει να αποφεύγουμε επίσης για την κατάτμιση των πληροφοριών, των δεδομένων και φυσικά η μη συμμετοχή σε μια τέτοια συνεργασία είναι έχει τραγικά αποτελέσματα και ξέρουμε πολλές τέτοιε περιπτώσεις στη χώρα μας. Τέλος πάντων τώρα το θέμα είναι η εποπτεία και ο έλεγχο από πλευρά των κοινοβουλίων ακριβώς ε, όπως ε, είπαμε ότι θα λειτουργήσει ούτω ώστε να υπάρχει περισσότερη νομιμοποίηση, να υπάρχει ε, λογοδοσία και θα πρέπει να υπάρχει μόνο ο έλεγχο και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωριστά και σε συνεργασία. Το θέμα δεν είναι επομένω να κάνει κανεί μια μεγάλη συνέλευση, μια μεγάλη διάσκεψη για αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο εισηγητή ο κ. Ντεμέρα, ότι θα πρέπει να θα έχουμε απλώ αυτή την ελεγκτική ομάδα. Και να δούμε ότι αυτό το σύστημα θα είναι πιο ελαφρό, πιο ευέλικτο, πιο λειτουργικό. Δηλαδή, Βεβαίω θα πρέπει να έχει όλη το σχετικό υλικό, την τεκμηρίωση. Όχι να ανακατεύεται στα εμπιέσεις της Europol, αλλά ότι θα ενημερώνεται ενημερώνεται με λειτουργικό τρόπο. Οπότε έτσι αν προσπαθήσουμε τότε θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στο να αποκτήσει περισσότερη ασφαλή Ευρώπη αλλά ίσως ο υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε κύριε Μωρένο, λέει ο πρόεδρο και τώρα. Ευρωβουλευτή. Κύριε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα και εγώ σύντομη θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα. Πρώτα απ' όλα η ομάδα μας τον υποστηρίζει ξεκάθαρα όσον αφορά το θέμα σε Πολ και τον διαχωρισμό τους. Δεύτερον, θα θέλαμε να συμπεριληφθούν και οι εθνικοί επόπτες δεδομένων και όχι μόνο ο Ευρωπαίος όσον αφορά την εποπτεία της Ευρωπόλ. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το τρίτον, βεβαίω ε, είμαι υπέρ του θεσμικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αναφέρθηκε μια επιτροπή κοινοβουλευτική ελέγχου όπως έχουμε στην ε, Γερμανία. Αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σωστό και βλέπουμε πως η διαφάνεια στην Ευρωπόλ τίνει προς το μηδέν και αυτό πρέπει να αλλάξει και τέλος ε, για το θέμα της ε, προστασίας των δεδομένων θα πρέπει νομίζω οι εκπροσώποι των, του Κοινοβουλίου να καθίσουν μαζί με τον κύριο Τίας Δεμέρα για να δούμε και στην ε, πράξη πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Νομίζω γενικά λοιπόν πως είμαστε σε καλό δρόμο και χαίρομαι για τις ε, προτάσεις του κυρίου Δίας Δεμερά. Ε, κρίμα που έφυγε αλλά θα του τα μεταφέρω ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ρέκορτ τώρα από τις κάτω χώρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προλαλήσαντες για την εισαγωγή και έχω κάποιες πρακτικές ερωτήσεις. Ε, μιλάμε για δημοκρατικό έλεγχο, ακούστηκαν πολλά και ε, εμένα με ενδιαφέρουν οι πληροφορίες που δεν μπορούν να είναι δημόσιες. Η αστυνομία εργάζεται και με απόρριτες πληροφορίες. Βεβαίως το ερώτημα απευθυνόταν στον κύριο Δίας Δεμέρα, αλλά απευθύνεται και στον κύριο Νόημαν, μια που είναι εδώ. Μπορεί λοιπόν να μας εξηγήσει ο κύριος ε, Νόημαν πώς θα υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος ε, με τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Εμείς ε, στην Ολλανδία έχουμε μια συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών όπου ενημερώνονται οι, προ... οι των κοινοβουλευτικών ομάδων για τα απόρριτα. Αν δεν γίνεται αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον δημοκρατικό έλεγχο. Αυτή ήταν η ερώτησή μου κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριο Σκαβλίδης από την Κύπρο. Ήθελα να ρωτήσω αν σκεφτήκατε καθόλου να συμπεριλάβετε σαν αρμοδιότητα του συντονιστικού οργάνου που θα ελέγχει τη Europol την εξέταση παραπώνων των πολιτών για κατάχρηση κατά την άσκηση των επιχειρήσεων. Αυτό παίρνει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας του διαδικτυακού εγκλήματος, παιδικής πορνογραφίας και άλλα, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Τα εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν οι πληροφορίες που τους διαβιβάστηκαν από τη Europol, είτε αυτές λήφθηκαν από την ίδια, είτε προέρχονται από κράτη-μέλη. Και έχουν τον κίνδυνο πολλές φορές να καταδικάζουν άτομα βασισμένοι σε μαρτυρία που προέρχεται από fruits of a poisonous tree. Γι' αυτό θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε το θέμα της άσκησης ενός προληπτικού ελέγχου όταν πολίτες που τίθενται υπό εκφράζουν κάποια παράπονα προτού τα στοιχεία ε, ληφθούν υπόψη από τα δικαστήρια. Δηλαδή στο στάδιο που θα διαβιβαστούν ε, θα τεθούν υπόψη των κατηγορουμένων και πριν γίνει η εκδίκαση της υπόθεσής τους. Ευχαριστώ. Now for Κύριος Μπρόνς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπόλ περιορίζεται στην υποψία διάπραξη σοβαρών αδικημάτων ή εμπλέκεται και σε παρακολούθηση δραστηριοτήτων, ειδικά πολιτικών δραστηριοτήτων που δεν είναι ποινικά αδικήματα. Όσον αφορά τα αδικήματα, πόσο σοβαρά πρέπει να είναι για να απασχολήσουν την Ευρωπόλ. Εκεί όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών για τον ορισμό ή ακόμα και το αξιόπινο κάποιας πράξης, τότε ένα κράτος μέλος και η αστυνομία του θα πρέπει να δώσει πληροφορίες για μια δραστηριότητα η οποία δεν είναι αξιόπινη στη χώρα αυτή. Αντιλαμβάνομαι επίσης πως ε, οι προτινόμενες ε, εποπτικές αρχές δεν μπορούν να εποπτεύσουν ε, τις επιχειρήσεις. Ε, μπορούν όμως να, να τις παρακολουθούν για να αντλήσουν κάποια γενικά συμπεράσματα. Εάν η Ευρωπόλ υπερβεί τις αρμοδιότητές της, τι μπορούν να κάνουν οι υφιστάμενες και προτινόμενες εποπτικές αρχές. Μπορούν να ξεκινήσουν μία έρευνα και πειθαρχικές διαδικασίες. Αυτά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας, ε, για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Λίγα λεπτά τώρα για τα μέλη του πάνελ να κάνουν κάποια σχόλια πριν ε, ακούσουμε την παρουσίαση των κυριών Λεμπάγι και Μάλστον. Λόρδε Χανί. Δεν θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις γιατί δεν υπάρχει και χρόνος. Αλλά μου έκανε εντύπωση το ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ε, σύγκληση στην στήριξη της πρότασης της ε, Κομισιόν και αυτά τα οποία ακούστηκαν ε, είναι βεβαίως πάρα πολύ σοβαρά αλλά δεν αφισβητούν την βάση. Κάποια πράγματα τώρα. Η Βρετανία είναι πολύ περισσότερο μια χώρα προορισμού και όχι διέλευσης για την παράνομη μετανάστευση, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες διέλευσης για, να μην υπάρξει αύξηση στην παράνομη μετανάστευση ε, από την οποία υποφέρουμε. Και νομίζω πως ε, η οδηγία περί τράφικινγκ που υιοθετήθηκε προσφάτως νομίζω πως θα είναι χρήσιμη. Κατόπιν, το θέμα των ε, καταγγελιών που ανέφερε ο βουλευτής από την Κύπρο. Βεβαίω ένα από τα αποτελέσματα του νέου κανονισμού όταν τεθεί ενισχύ είναι πως ε, θα προβλέπει την ε, υποχρεωτική δικαιοδοσία του ΔΕΚ, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτι το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή για την Ευρωπόλα και το έχουν δεχτεί εθελοντικά κάποια κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανική κυβέρνηση για να κρίνει αν θα ενταχθεί ή όχι σε αυτά τα μέτρα. Αλλά νομίζω πως θα απαντηθεί εν μέρει έτσι το ερώτημα που ετέθη. Φαίνεται πως η συγχώνευση του ΣΥΠΟΛ και της Ευρωπόλ ε, δεν ε, είναι πολύ δημοφιλής και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Τώρα για τις θεσμικές δομές της εποπτείας. Είναι σαφές πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι το πολύ λεπτομερές και χρονοβόρο και ακριβό. Και θα είναι λάθος αυτό. Ε, υπήρξαν κάποιες χρήσιμες ε, συζητήσεις ε, μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων και συμμετείχα και εγώ. Και αυτό το οποίο προέκυψε από την πρόταση της Κομισιόν είναι νομίζω πως πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Ελπίζω πως δεν θα το παραφορτώσουμε στην ε, διαπραγμάτευση με ζητήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα και πάνω απ' όλα έχει σημασία να μην μπούμε εμείς στην επιχειρησιακή λειτουργία της αστυνομίας. Δεν γίνεται αυτό στις χώρες μας και δεν πρέπει να γίνει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς θα έχουμε ε, μια λιγότερο αποτελεσματική αστυνομία. Τέλος, τα στατιστικά στοιχεία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τα λόγια να κοιτάμε και τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης της Ευρωπόλ, των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μέσων συνεργασίας. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει αύξηση της ε, χρήσης ε, της διαδικασίας αυτής στην Χάγη και αυτό νομίζω είναι η καλύτερη απόδειξη της ε, πραγματικής, πραγματικής της αξίας. Ευχαριστούμε Λόρθα Χάνη για το ότι ήσασταν και σύντομος. Κάποια άλλα σχόλια ίσως από τον κύριο Χάστινγκς, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ναι, δύο πράγματα. Άκουσα κάποια σχόλια που έλεγαν πως είναι σημαντική η προστασία δεδομένων, αλλά δεν πρέπει να αποθαρρύνει την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των εθνικών διοκτικών αρχών. Σύμφωνο, υπό την αίρεση πως είναι ε, σωστές, η σωστή ανταλλαγή πληροφοριών αυτή η οποία γίνεται. Και η πρόταση που έχουμε μπροστά μας θα την διευκολύνει, αλλά θα συμπεριλάβει κάποιες δικλίδες ασφαλείας ακριβώς για να ξέρουμε πως είναι ε, η σωστή και κατάλληλη ανταλλαγή η οποία γίνεται. Υπάρχει μια ισορροπία αυτή τη στιγμή και πρέπει να υπάρχει και στο μέλλον. Κατόπιν για την προτινόμενη δομή εποπτείας τόνισα την ανάγκη μιας συνολικής άποψης ε, που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ε, πτυχές και πρέπει νομίζω να υπάρχει και μια σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων. Η δομή που έχουμε τώρα ε, ε, έχει, από, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990, έχει λίγες αρμοδιότητες και περιορισμένη ανεξαρτησία και η προτινόμενη δομή οπωσδήποτε θα συμπεριλάβει τους εθνικούς επόπτες δεδομένων στο, πλαίσιο της εντολής τους. Π.χ. εάν μιλάμε για αυξημένη συνεργασία των εθνικών μονάδων εντός της Europol, εδώ πέρα υπάρχει αρμοδιότητα των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων. Αλλά μην μπερδευόμαστε. Εάν δοθούν εξουσίες εποπτείας στην ίδια τη Europol, ε, σε μια συνεδρίαση, τότε δεν είναι σαφής αυτή η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Οπότε εγώ θα ήθελα μια εποπτεία στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας. Αλλά α, πρέπει βεβαίως να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα από εδώ και μπρος και σύμφωνα με ευρωπαϊκά κριτήρια. Σας ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος Νόιμαν που εκπροσωπεί την Europol. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ με τα σχόλια του κ. Χάστινγκς ότι στον τομέα της Europol υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνεργασία. Όλο και πιο θετικά σχόλια ακούμε για τη δουλειά μας. Σας είμαι ευγνώμων και το θέμα της κοινοβουλευτικής εποπτείας και ελέγχου. Μπορούμε να αυξήσουμε την νομιμότητά μας και την εκτίμηση που χαίρει η δουλειά μας αν συνεργαζόμαστε με εμπιστοσύνη με το Κοινοβούλιο και αν μας ασκεί έλεγχο. Ε, σε ό,τι αφορά τα σχόλια του Ολλανδού βουλευτή, μπορώ να του πω ότι το σχέδιο κανονισμού της Europol ακριβώς αυτό προβλέπει. Προβλέπει να δημιουργηθεί δυνατότητα να γίνεται αυτή η πρόσβαση ε, και κλεισμένο των θυρών σε διαβαθμισμένες πληροφορίες οι εμπιστευτικές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του Βρετανού βουλευτή, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε απορρέουν από τα κράτη-μέλη στο μεγαλύτερο βαθμό και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε συλλέγονται από τα κράτη-μέλη νομίμως και έχουν ελεγχθεί από τα κράτη-μέλη πριν σταλούν στην Europol. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στις βάσεις δεδομένων μας είναι πληροφορίες που εμπίπτουν στην εντολή μας και δεν είναι εκτός αυτής. Έτσι ολοκληρώνω την τις απαντήσεις μου. Σας ευχαριστώ όλους, όλους τους πήρατε το λόγο και τους εθνικούς βουλευτές και τους ευρωβουλευτές. Και τώρα η κυρία Φρανσουάς Λεμπάι, που είναι Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ε, Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την καλωσορίζουμε για το δεύτερο τμήμα αυτής της συζήτησης. Η κατάσταση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποινικέ υποθέσεις. Έχετε το λόγο, κυρία Λεμπάγη. Thanks again for Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, θα ακούσουμε την παρουσίαση της κυρίας Λεμπάγια για το θέμα που προανέφερα και αν έρθει στο μεταξύ και η, Επίτροπη, και η Επίτροπος Μάλστρομ Θα ακούσουμε διάφορες ερωτήσεις από το κοινό προς την ε, Γενική Διευθύντρια και την Επίτροπο. Κυρία Λεμπάγη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ε, εφαρμογή του προγράμματος Χόλμης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θέτει τους Ευρωπαίους πολίτες στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Κομισιόν που ανέλαβε τα, τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 2010 έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, ούτω ώστε αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης να γίνει μια πραγματικότητα. Είναι σημαντικό αυτό, σε αυτή τη φάση τώρα, να σταματήσουμε λίγο και να δούμε τα πράγματα από μια απόσταση, να δούμε πού φτάσαμε σε αυτή τη ε, φάση της εφαρμογής και να το κάνουμε όχι μόνο με, τα με τους φίλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά να έχουμε κάποια στιγμή και την ευκαιρία να το κάνουμε με τους εθνικούς βουλευτές, που παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο επίπεδο αυτό. Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στα εθνικά κοινοβούλια ένα ρόλο. Και χάρη σε αυτά η αρχή της επικουρικότητας, φερρυπίν μεταξύ άλλων, γίνεται σεβαστή. Σε ένα τομέα που είναι τόσο κοντά στη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών όπως είναι η δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ηθαγένεια, το, τα εθνικά κοινοβούλια παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το Ευρωκοινοβούλιο φυσικά. Θέλω λοιπόν τώρα να διατρέξουμε μαζί όλα τα επιτεύγματα που υλοποιήσαμε και όλες τις πολιτικές που εντάσσονται και απορρέουν από το πρόγραμμα της, Λισαβο, της Στοκχόλμης. Θα σας μιλήσω για τις ε, πρωτοβουλίες στον τομέα του ποινικού δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Αυτά καλύπτει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης στο δικό μου τομέα. Ας ξεκινήσουμε με, τους πολίτες. Γιατί εδώ μιλάμε με εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων σήμερα και νομίζω ότι ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα του προγράμματος της Στοκχόλμης είναι ότι θέτει τους πολίτες στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης. Σε αυτό τον συγκεκριμένο τομέα παρουσιάσαμε μια νέα έκθεση για την ηθαγένεια που είναι ένας πρακτικός τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι η ζωή των πολιτών θα βελτιωθεί. Επίσης, υποβάλαμε μία έκθεση, ετήσια είναι αυτή, για τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο στόχος της δεν ήταν να απλώς να τη γράψουμε, αλλά να δείξουμε τι πρόοδο έχουμε σημειώσει στην εφαρμογή της χάρτας. Και πώς η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει απλουστευτεί και έχει οδηγήσει και καθοδηγήσει τις βασικές πολιτικές των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Και επίσης ψάξαμε να δούμε και τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στα κράτη-μέλη. Καταρχάς, με μεγάλη έμφαση πολεμήσαμε για την ισότητα άνδρων και γυναικών. Η Κομισιόν έκανε μία πρόταση για τις ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια εταιριών. Μία πρόταση η οποία ήταν πολύ αμφιλεγόμενη. Ακούστηκαν πολλές επικρίσεις. Αλλά η πρόταση αυτή ήταν και μία απεικόνηση της επιθυμίας μας να υπάρξει ισότητα στα διοικητικά συμβούλια των ε, εταιριών. Επομένως, θέτουμε πραγματικά τους πολίτες στο κέντρο της δράσης μας και ένα από τα θέματα που προωθήσαμε και νομίζω ότι ο Πίτερ Χέστινγκς το ανέφερε προηγουμένως, είναι η προστασία των δεδομένων. Για την προστασία των δεδομένων αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών γιατί όλοι μας όλο και περισσότερο μέσω της χρήσης του ίντερνετ δίνουμε τα δεδομένα μας. Και επομένως είναι και η ώρα να προσαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία σε αυτές τις νέες απαιτήσει της τεχνολογίας. Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας ακριβώς, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για θέματα προστασίας των δεδομένων. Και ακριβώ για αυτό το θέμα είμαστε σε συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μεταρρύθμιση τη προστασία των δεδομένων συνδέεται και με την ε, ενίσχυση του δικαιώματο των πολιτών και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ευρωπαϊκών εταιριών. Θέλουμε να ενισχύσουμε ε, ένα κοινό καθεστώς προστασίας των δεδομένων παρά 27 ε, διαφορετικών. Πιστεύουμε ότι εδώ θα έχουμε εξοικονόμηση πάνω από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο χάρη σε αυτή την προσπάθεια. Βάζουμε τους πολίτες στην καρδιά, ενισχύουμε τα δικαιώματά τους έτσι λοιπόν και εξασφαλίσουμε ότι η δράση μας στον τομέα της δικαιοσύνης συνδέεται και με την ανάπτυξη. Σε σχέση με την ανάπτυξη επίσης, η σημερινή Κομισιόν πρότεινε και μέτρα όπως η εξάλληψη του, της εκτελεστότητας, του εκτελεστού τίτλου, του εξεκουατούρ. Ε, α, το εξεκουάτουρ ε, κοστίζει 48 εκατομμύρια το χρόνο χωρίς κανένα λόγο. Ε, το απλουστεύσαμε λοιπόν. Επίσης κάναμε προστα... προτάσεις για την αφαιρεγκαιότητα. Ο σκοπός αυτών των προτάσεων είναι να εξασφαλίσουμε ότι όταν μια εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία. Και τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της εταιρείας, αν ας πούμε οι δυσκολίες είναι μόνο προσωρινές, όλα ελέγχονται, ούτως ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην επιβίωση της εταιρείας. Αυτό λοιπόν είναι τμήμα της δράσης μας και συνδέεται προφανώς με την ανάπτυξη. Επίσης, κάναμε μια πρόταση για το εταιρικό δίκαιο, για το δίκαιο των συμβάσεων, συγγνώμη. Επίσης για τις μικρές απαιτήσει, ούτω ώστε οι καταναλωτές και οι εταιρείε να παίρνουν γρήγορα τα λεφτά τους πίσω. Ε, απλουστεύουμε τις διαδικασίες Θέλουμε να τις απλουστεύσουμε περαιτέρω και πιστεύουμε ότι το όριο που είχαμε μέχρι στιγμής για τις μικρές απαιτήσει, που ήταν 2.000, είναι πολύ μικρό. Και θέλουμε να αυξήσουμε αυτό το όριο, να μιλήσουμε για απαιτήσει μέχρι δηλαδή 10.000 οικονομικές αξιώσεις, μέχρι 10.000. Είναι ε, μέτρα για την δικαιοσύνη και την ανάπτυξη πολύ σημαντικά. Στη δράση που παρουσιάσαμε και υιοθετήσαμε υπάρχουν επίσης μέτρα προς όφελος των οικογενειών. Φερρυπίν. Εισάγουμε νέους κανόνες, τους εισήγαμε το 2010, για τις διαδικασίες διαζυγίου, για ζευγάρια μικτά από διαφορετικές χώρες. Το 2004 είχαμε πάνω από 100.000 τέτοια ζευγάρια και γι' αυτό οι διαδικασίες θα απλουστευτούν πάρα πολύ. Επίσης κάνω μια πρόταση για, την... για το διακανονισμό διεθνών κληρονομιών. Θέλουμε να υπάρχει ξεκάθαρο δίκαιο, σαφής δικαιοδοσία Όταν υπάρχουν κληρονομιές με διεθνή διάσταση, ε, ύψους πάνω από 450.000 ευρώ. Θέλουμε έτσι να αυξήσουμε την καθημερινότητα των οικογενειών. Στο ποινικό δίκαιο έχουμε πετύχει πάρα πολλά με την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων. Είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις και επί Βελγικής Προεδρίας για την πρόσβαση σε δικηγόρο, Φερρυπίν. Αλλά και το δικαίωμα σε διερμηνία, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αν σε συλλάβουν, Φερρυπίν, σε ένα κρατός μέλος, θα έχεις κάποια ελάχιστα δικαιώματα, τα οποία θα σε προστατεύουν, αν είσαι ύποπτος. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Η πρόταση για πρόσβαση σε δικηγόρο, κατά την απόψή μας, είναι πολύ σημαντική στον τομέα του δικονομικού δικαίου. Προσπαθήσαμε να έχουμε μία μακρόπνοη θεώρηση. Ο προβληματισμός που ξεκινήσαμε για τη δημιουργία Ευρωπαίων εισαγγελέων την επόμενη, στην επόμενη σύνοδο θα έχετε την ευκαιρία να το συζητήσετε αυτό το θέμα πιο λεπτομερώς. Αλλά η ιδέα πίσω από τη δημιουργία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που θα προτείνει η Κομισιόν σύντομα πιστεύω, θα ενισχύσει τον αγώνα κατά του εγκλήματος και την επίθεση εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτή η ιδέα, η προστασία των οικονομικών συμφερόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία των πολιτών, αυτή η ιδέα διαπερνά όλες μας τις πολιτικές και προτάσεις. Και νομίζω ότι χάρη σε όλες αυτές τις προτάσεις μπορούμε να συνεισφέρουμε και στην ανάπτυξη. Αυτές οι, αυτά τα επιτεύγματα δεν ήταν πάντα εύκολα να σημειωθούν. βρίσκονται στην καρδιά της πολιτικής μας για τη δικαιοσύνη, των παραδόσεων για τη δικαιοσύνη, για τη δικαιοσύνη των αξιών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Και εκεί έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, πιστεύω. Υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη, το Justice Scoreboard. Θέλουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα δικαστικά μας συστήματα για την πρόθεση της ανάπτυξης, για την προστασία των πολιτών. Φερρυπίν, αν είσαι μια επιχείρηση, πόσο χρόνο χρειάζεται για να πετύχεις μια απόφαση, πόσο κοστίζει κτλ. κτλ. Ήταν μια πρώτη απόπειρα αυτό το, αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων. Αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα και δείχνουν πραγματικά το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η δικαιοσύνη σε κάποια, άλλα κράτη, σε κάποια κράτη-μέλη και πόσες καθυστερήσεις ας πούμε, παρουσιάζουν κάποια άλλα. Έχουμε βάλει στους πίνακες ε, νούμερα, αριθμητικά στοιχεία και φυσικά ευθύνη της δράσης σε αυτό το επίπεδο είναι εμπίπτει στα κράτη-μέλη. Αλλά μας δείχνει ακριβώς την ε, πρόοδο που έχει σημειωθεί και αυτό δημιουργεί μια εμπιστοσύνη σε επενδυτές να έρθουν εδώ, να εγκατασταθούν σε κράτη-μέλη, να επενδύσουν. Γιατί ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα είναι συνιστόσα της ανάπτυξης και της ανάκαμψης. Αυτά σε δύο λόγια τα είπα. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά ο Πρόεδρος θα δυσανασχετούσε. Όλα αυτά σας δείχνουν πόσα πράγματα πετύχαμε σε αυτόν τον τομέα. Τώρα βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Το κάνει το Κοινοβούλιο σε μια έκθεση και εμεί το σκεφτόμαστε αυτό το θέμα. Θα γίνει το Νοέμβριο μια μεγάλη α, διάσκεψη, les assises de la justice όπως λέμε στα γαλλικά, η διάσκεψη για τη δικαιοσύνη και θα προβληματιστούμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμεί σα ευχαριστούμε για όσο μα παρουσιάσετε από πλευρά Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, για το χαρτοφυλάκιό σα. Πάντω, ε, Χθε είχε έρθει εδώ η Επιτροπός Ρέντιν και μας είπε για αυτό το συμπόσιο για θέματα δικαιοσύνης το οποίο θα οργανώσετε. Πάντως, ε, οπωσδήποτε, ε, και σήμερα έχουμε την Επίτροπο Μάλμστρομ θα τιμήσει την συνάντησή μας. Ε, είναι Επίτροπος Ιστορικών Υποθέσεων. Και με την Επίτροπο θα ολοκληρώσει αυτό το τμήμα της ημερίδας μας. Και μετά από την κυρία μας θα αρχίσει η συζήτηση με τους ε, βουλευτές με την ίδια διαδικασία. About the fields of subject matter that are being discussed. Commissioner Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι εθνικοί βουλευτές και βουλευτές του Κοινοβουλίου, κυρία Διευθύντρια. Μεγάλη μου τιμή και εγώ έρχομαι σήμερα στο συνάντησή σας για το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Το 2009 ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, η οποία τώρα όπου να θα ολοκληρωθεί. Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε μια γενική αξιολόγηση και να σας πω για τα δικά μου θέματα τι πρόοδο έχουμε σημειώσει. Έχουμε ασπίσει μια σημαντική οδηγία για τη διακίνηση ανθρώπων, ούτως ώστε να μπορέσουμε ε, αυτή την ε, πληγή της εποχής να την ε, εκριζώσουμε και με τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο επίσης. Έχουμε μια πρωτοβουλία για την εκμετάλλευση των ανηλίκων, την σεξουαλική προστασία των, των, των θυμάτων δίωξη κατά των υπευθύνων. Επίσης έχουμε μια οδηγία για τα πυροβολά όπλα και ε, επίσης ε, για τα στοιχεία επιβατών αεροπλάνων, το PNR, έχουμε συνεργασία με ΙΠΑ, Αυστραλία και Καναδά και επίσης ε, θέλουμε να υπάρξει ένα ένα δίκτυο το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και με αυτό το δίκτυο θέλουμε να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε όλα τα επίπεδα για όλα αυτά τα, για τα φαινόμενα ε, της ε, παστικοποίησης δηλαδή το, το πώς κάποιοι ε, εξωθούνται κατόπιν κατόπιν κάποιας κατήχησης να κάνουν βίες πράξεις. Και οπότε θα θυμάστε ότι είχαμε πάρα πολύ ευρία πλειοψηφία για τις οδηγίες όσον αφορά την διαδικασία χορηγής ασύλου. Τα κρατημελή βεβαίως έχουν αναπτύξει μια δραστηριότητα σημαντική, οπότε και τώρα έχουμε πιο συνεπή ε, πολιτική, πιο καλή διαδικασία για εκείνους ε, οι οποίοι αναζητούν ε, άσυλο, αναζητούν καταφύγιο στα κράτη-μέλη. Επίσης έχουμε κάποια μέτρα όσον αφορά την περιοχή Σέγγεν. Αυτό δεν είναι το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Όμως χρειαζόντουσαν αυτά τα μέτρα και βλέπετε το ότι απαιτείται ευελιξία και στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Δεν πρέπει δηλαδή κανεί να κολλάει σε ένα πρόγραμμα πενταετέ γιατί τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Πάντω έχουμε κάποιε σημαντικέ ε, νομοθετικέ προτάσει, έχουμε κάποια νομοθετήματα που συζητούνται, δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Η κυρία Λουμπάη σα είπε για την καταπολέμηση του εγκλήματο και εμεί συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια γιατί βεβαίω ε, πρέπει να δούμε ότι θίγονται τα θύματα, θίγεται η κοινωνία, αλλά έχουμε και την οικονομική επιτυχία γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σχετίζονται με το έγκλημα. Οπότε και εμείς θέλουμε να υπάρχει ανάκτηση αυτών των ε, χρημάτων και να επιστρέφονται στους φορολογουμένους. Έχουμε το θέμα της κατάσχεσης των προϊόντων εγκλήματος και κατά τρόπο νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι αντικίνητρο οικονομικό για το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, το φθινόπωρο θα έχουμε την πρώτη έκθεση κατά της διαφθοράς. Θα τονίσουμε τι πάει καλά στα κράτη-μέλη, αλλά θα πούμε και το τι χρειάζεται να κάνουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την διαφορά που υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Και επίσης 120 δις θεωρείται το κόστος αυτό της ε, διαφθοράς. Οπότε για φανταστείτε Οπότε, ε, να ρίξουμε τώρα και μία ματιά στις προοπτικές στο μέλλον, τι γίνεται με τις νίκη της Λισαβόνας, γιατί τα εσωτερικά τώρα πια είναι ε, κάτι το οποίο δεν είναι διακυβερνητικό, κάτι το οποίο θα διευνεί όλες τις πολιτικές της κοινότητας. Έχουμε επομένω ε, την ιδιότητα του συνομοθέτη τώρα με συμβούλιο και κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσέγγιση, θα πρέπει να έχουμε ε, ένα ενδελεχές ε, πρόγραμμα και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης επίσης ε, σχετίζεται με αυτή την καινούργια κατάσταση, η αναβάθμιση Εθνικών Κοινοβουλίων, αναβάθμιση προβλέπεται και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις νέες σας αρμοδιότητες. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και, τα θέματα υλοποίηση, να δούμε όμως και τις προτεραιότητες. Θα συνεννοηθούμε μαζί σας, θα συντονιστούμε με τα κρατημέλη, με πανεπιστημιακούς, με κυβερνητικούς οργανισμούς και έτσι θα υπάρξει για την αυριανή πολιτική ένας ε, δυναμικός διάλογος. Έχουμε επίσης και ε, το άτυπο συμβούλιο υπουργών εσωτερικών που θα γίνει στην Λιθουανία σε ε, λίγες εβδομάδες. Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι τώρα οι κοινέ προκλήσεις πώς θα προστατευτεί ο πολίτης, οι νέες απειλές, τρομοκρατία, κυβερνοέγκλημα, διακίνηση ανθρώπων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πώς θα έχουμε περισσότερη ελληνική, πώς θα έχουμε εφαρμογή του νόμου, πώς θα εξασφαλίσουμε ε, το να είναι η Ευρώπη ασφαλής περιοχή, αλλά και πώς θα ανακτήσουμε το τα προϊόντα, τα χρήματα που βγαίνουν από το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε και έτσι θα προσπαθήσουμε να υπάρχει σεβασμός περισσότερων ανθρώπινων δικαιώματων εκτός από το να είναι η Ευρώπη ασφαλής και ασφαλέστερη. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο για την Europol, γιατί ξέρω ότι είναι το θέμα της σημερινής σας ε, ε, συνάντησης. Ε, να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα είναι η Europol, την άμεση της Λισαβόνας. Θέλουμε μια καλύτερη Europol, καλύτερα πληροφορημένη, να συμβολεί καλύτερα στη συλλογή πληροφοριών, να έχουμε την διαχείριση των δεδομένων πιο ευέλικτη, να έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών και επίσης να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Θέλουμε να υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχος. Για πρώτη φορά θα εμπλακούν εδώ και τα εθνικά κοινοβούλια. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε αποδοση ευθυνών, πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες και ε, εσείς ξέρετε πώς θα συνεργαστείτε, αλλά Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για να μπορέσει να υλοποιήσει την εντολή της η Europol για να είναι πιο αποτελεσματική και ακολουθώντας του προβλεπόμενους κανόνες και στη διοίκηση και στα οικονομικά. Έχουμε διαφορετικές προτάσεις να σας παρουσιάσουμε, έτσι εσείς νομίζω ότι κάνετε τον έλεγχό σας και διαβούλευση για το πολιετές πρόγραμμα, ε, για τις απειλές, για τις δραστηριότητες, εκθέσεις. Ε, θα έχει να έχετε επίσης τον ετήσιο προγραμματισμό και να συνεχίσετε βέβαια τον ρόλο σας σαν αρχή του προπολογισμού για διοικητικό συμβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο ε, και επίσης όλα αυτά θα συζητώνται και σε συναντήσεις όπως η σημερινή και θα υπάρχει και κάποιο είδους ε, κατάρτιση, εκπαίδευση για την εφαρμογή του νόμου που θα είναι στην καρδιά του συστήματος. Ίσως ήδη εσείς ξέρετε τις προτάσεις Κομισιόν για τη συγχώνευση Europol και Σεπόλ. Νομίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερη συνέργεια, έτσι θα απελευθερώσουμε κάποιους πόρους για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα της κατάρτισης και θα βοηθήσουμε τώρα για κάποιες καινούργιες υπηρεσίες. Επίση, ε, είπαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κλείσει το Μπράμσελ, οπότε η εκπαίδευση θα γίνεται στη Χάγη, στην Europol. Εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε οικονομίες, θα πρέπει να βρούμε από αλλού το, τα χρήματα που χρειάζονται. Βέβαια έχουμε το, το, το ε, πρόγραμμα, οπότε αν θέλουμε να κάνουμε την κατάρτιση που είπαμε πρέπει να ξεβρεθούν τα χρήματα γι' αυτό και ήρθαμε εδώ με την Φρανσουάζ και θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Είμαι βέβαιη ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, θα υπάρχει συνέχεια για το ποιες θα είναι οι γραμμές στην πολιτική μας ε, για το μέλλον. Εμείς ευχαριστούμε κυρία μου λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και την Γενική Διευθύντρια για την εισήγησή Μα γι' αυτό ακριβώς και ε, θέλουμε να υπάρχει αυτό το διακοινοβουλευτικό βήμα. Προβλέπονται αυτά ώστε από τις συνήθειες και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εμπλέκει όχι μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά και τα κοινοβούλια. Για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Μιλήσατε και για την Europol. Γιατί υπάρχει το ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί. Θα γίνει αυτή η συγχώνευση. Τα είπαμε και στην αρχή της ε, σημερινής ημερίδας, αλλά πάντως τώρα τη σκητάλη θα έχουν οι βουλευτές για παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πρώτος, σύμφωνα με τον κατάλογο, αυτό μου ζητήσει το λόγο, θα μιλήσει ο κύριος Φάλσον από το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε σε ένα πράγμα πως έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία, όπως είπε και η Επίτροπος κυρία Μάλστρομ, ειδικά η διασυνοριακή φύση του εγκλήματος όπως η εμπορία ανθρώπων, ε, όπλων, ναρκωτικών ε, κτλ. Επειδή είμαι Μαλτέζος, ε, λογικό είναι να πω κάτι για την λαθρομετανάστευση και η κυρία Μάλμστρομ αναφέρθηκε σε αλλαγές και βελτιώσεις στην διαδικασία ασύλου κατά το οποίο έχει δημιουργήσει συζητήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα καλά, αυτά, οι προδιαγραφές ε, και τα σχετικά, αλλά τι θα γίνει και με τις ε, συνθήκες ε, στις χώρες υποδοχής όπως η δική μου. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η Μάλτα είναι η 8η χώρα στον κόσμο, μιλάμε τώρα για χώρες μαζί με την Ιορδανία όπου ξέρουμε που έχει οδηγηθεί η κατάσταση, και υψηλότερη στον κόσμο όσον αφορά την υποδοχή ανθρώπων. Ε, πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Ωραίο είναι αυτό να μιλάει κανείς από μακριά, έτσι, για τη βελτίωση προδιαγραφών και ε, όλοι συμφωνούμε βεβαίως, ε, συνεργασία όλοι συμφωνούμε, αλλά τα βάρη που επομίζονται κάποιες χώρες όπως η δική μου, που είναι κατά βάση στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου η συνεργασία με τις τρίτες χώρες εκτός Ένωσης ε, από όπου έρχεται η παράνομη μετανάστευση ή οι ετούντες άσυλο, γιατί συνέχεια αλλάζεται τις λέξεις, ε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνεργασία. Τι γίνεται εκεί. Σας ευχαριστώ. κύριο Σεβερίνσκι, πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ε, Πολωνική Γερουσία. Κύριε Σεβερίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για την πρόταση αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα από την Κομισιόν. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αυξανόμενη δραστηριότητα της Γεροπόλ και τις πολύτιμες υπηρεσίε της καθώς βοηθάει τα εθνικά θεσμικά όργανα. Η αυξανόμενη ροή δεδομένων είναι αναπόφευκτη και θα είναι στα χέρια των ε, οργάνων της Ευρωπόλ. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά μέσα ελέγχου και εποπτείας. Ειδικά για να προστατεύσουμε τα δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα. Οπότε για να γίνει αυτό πρέπει να οργανώσουμε τη σωστή εποπτεία από πλευράς εθνικών κοινοβουλίων. Νομίζω πως η καλύτερη λύση, όπως προτάθηκε ήδη από κάποιον Γερμανό συνάλφο, ήταν μία διακοινοβουλευτική επιτροπή, αντί για κάτι ευρωπαϊκό και δυσκίνητο όπως αυτό. Όσον αφορά τη συγχώνευση Europol και νομίζω πως πρέπει να αποφευχθεί. Γιατί? Όταν αποκτήσουν κάποια σημασία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν την τάση να μεταβάλλονται σε φορείς ε, εξουσίας αντί να βοηθούν και να συμβουλεύουν τους εθνικούς φορείς. Οπότε θα ήθελα να τονίσω πάλι το ότι ο έλεγχος των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να διασφαλιστεί με αυτή την Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Είναι καλή ιδέα αυτή. Σας ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Σατζεντίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ. Κυρία Μάλστρομ, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, Τάμπερε, Χάγη ήταν διακυβερνητικά και το ερώτημα είναι αν πρέπει να έχει αυτή τη μορφή και στο μέλλον ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να ρωτήσω τι θέλετε να έχετε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον ή να μην έχετε όσον αφορά την ε, δικαστική συνεργασία. Γιατί κάποια πράγματα δεν ρυθμίζονται τώρα π.χ. το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πώς μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι άλλο από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, γιατί για να είμαι ειλικρινής, φαντάζομαι πως και οι εθνικοί βουλευτές αναρωτιούνται τι πρέπει να γίνει ε, αν είναι να αποστείλουν πολίτες τους σε άλλη χώρα, αν ξέρουν ε, το ότι οι συνθήκες στις φυλακές δεν είναι ιδανικές ή ότι δεν υπάρχει νομική αρρωγή. Ε, οπότε η επεξεργασία ενός νέου προγράμματος Στοκχόλμης δεν υπαρχει νομικη αρρωγη οποτε η επεξεργασια ενος νεου προγραμματος χολμη δεν πρεπει να αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας και να έχουμε μια κάποια εναρμόνιση και κάτι περισσότερο από την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί νομίζω πως δεν μπορούμε πλέον να αποφύγουμε, όπως είπα, αυτή την ε, ελάχιστη εναρμόνιση. Θέλει κάποιος άλλος, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος τον λόγο, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις. Κύριε Λεμπάχη. Ή εσεί ότι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Να αντιδράσω στις τελευταίες, ερω... μάλλον στην τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι μου απευθύνεται. Συμφωνώ ότι πρέπει να, πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος βαθμός νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε δημιουργούμε ελάχιστα ας πούμε, πρότυπα δικονομικά. Ακριβώς για να συνεισφέρουμε στην εμπιστοσύνη στο σύστημα ο ένας του άλλου. Άρα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο βαθμό νομοθεσίας. για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη. Είναι μια διακυβερνητική απόφαση όντω. αλλά από το Δεκέμβριο του χρόνου η Κομισιόν θα έχει την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη να ανασκουμποθούν. Πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο βαθμό νομοθεσίας και παράλληλα όλα αυτά τα μέτρα που προωθούμε για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη που έχει το ένα κράτος μέλος στη δικαιοσύνη του άλλου. Επίσης, σε κάποια φάση θα μιλήσουμε για την κατάρτιση, που είναι κάτι διαφορετικό. Να σας πω ότι σκοπεύουμε να καταρτήσουμε τους μισούς επαγγελματίε σε όλη την Ευρώπη από σήμερα μέχρι το 2020 στον τομέα της δικαιοσύνης. Επομένως, θέλουμε ελάχιστα πρότυπα, αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο συνδυασμό αυτών είναι η απάντηση για το μέλλον. Η Επίτροπος Μάλτρομ Με το ερώτημα του βουλευτή από τη Μάλτα. Είναι σημαντικό να έχουμε κοινού κανόνες και πρέπει να βοηθήσουμε όλες τις χώρες Φυσικά τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαφορετικές ε, γεωγραφικές θέσεις και καταλαβαίνω ότι οι χώρες όπως η Μάλτα ε, δέχονται πολλές ε, πιέσεις λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, αλλά και γιατί είναι πολύ μικρή χώρα και γιατί έχει μεγάλο πληθυσμό για την εκτασία της. Το ξέρουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις αρχές της Μάλτας όσο μπορούμε. Εγώ, ας πούμε, νεπλάκι στην δρομολόγηση του προγράμματος δεύτερης μετεγκατάστασης. Ε, όμως, 25 κράτη-μέλη ε, αρνήθηκαν το πρόγραμμα τη μόνιμη επανεγκατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τακτικό φόρουμ για να συζητάμε τέτοια θέματα, να αναλύουμε τι ροές και να δίνουμε έμφαση στι χώρε που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση. Σήμερα είναι η Μάλτα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι μια άλλη χώρα. Πολλέ χώρε εξάλλου, εκτό από τη Μάλτα και σήμερα αντιμετωπίζουν πολλέ πιέσει με τους κατάλληλους πόρους, χρήμα κτλ. Και, την, και τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε σε θελοντική βάση να εμπλέξουμε και άλλα κράτη-μέλη ε, να δεχθούν την επανεκατάσταση. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει. Αλλά ένα μόνιμο σύστημα αλληλεγγύης ή μετεγκατάστασης, αν θέλετε. Ξέρω ότι το, το θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν το θέλουν τα 25 από τα 27 κράτη-μέλη. Άρα τι να κάνουμε. Για την, τον έλεγχο της Europol, με ρώτησε κάποιος. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το πώς ε, οργανώνετε εσείς την συνεργασία σας δεν είναι δικό μου θέμα. Ξέρω θα το συζητήσετε περαιτέρω σήμερα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε εμπιστοσύνη να υπάρχει αυτή η συνεχής λογοδοσία και έλεγχος. Τώρα, για τις ΕΠΟΛ, Όλοι έχουν, όλα τα κρατημέλη έχουν φιλοδοξίες για τη ΣΕΠΟΛ σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και τη βελτίωση της αστυνομικής κουλτούρας και γνώσης σε όλη την Ευρώπη. Αλλά όμως με τις περικοπές που προβλέπουμε <laughs> δεν νομίζω ότι σήμερα ε, η ΣΕΠΟΛ μπορεί να τα καταφέρει. Γι' αυτό λοιπόν η συγχώνευση είναι μία λύση για να εξοικονομήσουμε πόρους. Τώρα, αν δεν συμφωνήσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την πρόταση, ακόμη και αν όλοι οι άλλοι έχουν συμφωνήσει, τότε θα πρέπει να ξαναδούμε όλες τις, ε, όλους τους οργανισμούς για να δούμε πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Μπορούμε να βρούμε από αλλού τις, ε, τα κονδύλια αυτά. Να δούμε πού αλλού μπορούμε να κάνουμε τις περικοπές. Το Κοινοβούλιο μπορεί να τα εξετάσει αυτά τα θέματα, μπορεί να τα συζητήσει και πέρα από τη συγχώνευση της ΕΠΟΛ με την ε, Europol μπορούμε συνολικά να δούμε την εικόνα χάρη στο Κοινοβούλιο γιατί χάρη σε αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λύση. Ε, για την ερώτηση της κυρίας Σαρτζεντίνη, γιατί δεν θέλουμε ένα κατάλογο. Κάποιες προτεραιότητες θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να εστιάσουμε σε αυτές, γι' αυτό ξεκινάμε αυτό το διάλογο. Ε, ακούμε αυτά που μας λέτε εσείς, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ένα λεπτομέρειο κατάλογο, γιατί αυτό ε, το κάναμε στις εποχές πριν της Λισαβόνας. Τώρα είναι συνήθις ε, τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής και δεν χρειάζονται αυτοί οι κατάλογοι. Αλλά βεβαίως κάποιες προτεραιότητες πρέπει να έχουμε και να τις συναποφασίσουμε μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ και τις δύο μιλήτριες, την κυρία Λεμπάιγε και την Επίτροπο Μάλστρομ. Αν μου επιτρέπετε και μένα τώρα, Να προσθέσω και εγώ κάτι ουσιαστικό. Όντως, παρακολουθούμε και αναλύουμε την κατάσταση του προγράμματος της Στοχόλμης, που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2009 επί Σουηδικής Προεδρίας. Ήταν το πρώτο μετά το πρόγραμμα Tampere το, του 1999 και μετά είχαμε το πρόγραμμα της Χάγης το 2004. Αυτά ίσχυαν πριν την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Τότε ίσχυε η δυναμική των κυβερνήσεων όπως εκπροσωπούνταν στο Συμβούλιο. Αυτές οι χώρες στο Συμβούλιο αποφάσιζαν τι θα γίνει στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με βάση τον, τα όσα ίσχυαν και τους κανόνες που ίσχυαν στον πρώην τρίτο πυλώνα. Τώρα όμως έχουμε να κάνουμε ευρωπαϊκές πολιτικές όπου εμπλέκονται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επομένως τα επόμενα πέντε χρόνια εάν κάποιο πρόγραμμα άλλο διαδεχθεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τα όσα λέει η Λισαβόνα τότε θα πρέπει να υπάρχει γι' αυτό μια διαθεσμική συμφωνία και βεβαίως θα πρέπει να εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα πρέπει το Συμβούλιο από μόνο του να αποφασίζει όπως συνέβαινε. Ακόμα και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μόνο του το αποφάσισε το Συμβούλιο, που το αποφάσισε στο τέλος του 2009 επί Σουηδικής Προεδρίας το Συμβούλιο. Τώρα όμως, όχι μόνο το Συμβούλιο, αλλά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουν. Τώρα έχουμε νέους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν έχουμε πια τη λεγόμενη διακυβερνητική συνεργασία. Ήθελα να το πω αυτό. Και επίσης κάτι άλλο που τονίζω πάντα είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση. Όχι μόνο των δικαστών και των εισαγγελέων, αλλά γενικά όσοι ασκούν το επάγγελμα, οι επαγγελματίες, δικηγόροι, σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να έχουν τη σωστή κατάρτιση, ούτω ώστε να εφαρμόσετε σωστά το ευρωπαϊκό δίκαιο στον τομέα που συζητάμε. Ούτω ώστε η δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει, να λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, που είναι τμήμα της συνθήκης Λισαβόνας. Επομένω, η κατάρτιση των νομομαθών είναι εκ των όνου Να μαθαίνουν το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά όχι μόνο, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να τους διδάξουμε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι αποτελεσματικό μόνο αν λάβουν υπόψη την προστιθέμενη αξία του οι επαγγελματίες. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε ένα νέο ε, πάνελ ομιλητών για την τελευταία μας ε, συζήτηση σήμερα το πρωί. We welcome in the podium. Ορίζουμε τώρα τους επόμενους ε, ομιλητές μας, το τελευταίο κομμάτι της πρωινής συνεδρίασης, που έχει θέμα ακριβώς την αποτελεσματικότερη συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις και περνάμε άρα στη Eurojust, το Ευρωπαϊκό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 η Eurojust ήταν ο προπομπός του, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 της ε, Συνθήκης Λισαβόνας. Έχει υπάρξει πρόοδο στα θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ των οποίων προστασία των θυμάτων σε ποινικέ υποθέσεις. Ε, υπάρχει αυτό στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ε, στο σχέδιο δράσης δηλαδή της Κομισιόν. Είχαμε σημαντική πρόοδο στον τομέα των δικονομικών δικαιωμάτων, συγκεκριμένα δηλαδή ε, διερμηνία, μετάφραση, δικαίωμα της ε, πληροφόρησης ε, που έχουν ήδη εγκριθεί και τώρα θα εγκρίνουμε στην Ολομέλεια το δικαίωμα της πρόσβασης σε δικηγόρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εδώ πέρα λοιπόν μια πραγματική ουσιαστική διαφορά για τους Ευρωπαίους πολίτες και οδεύουμε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, για να αξιολογήσουμε ακριβώς ε, την ε, Eurojust. Όπως προβλέπετε στο άρθρο 85 της συνθήκης ε, που προβλέπει, επιμένω, την Eurojust ως μια αφετηρία για να καταλήξουμε τελικά σε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία. Σας ακούσουμε τώρα τους ομιλητές μας, μεταξύ των οποίων την κυρία Μαριέτα Κάραμανλή, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Καλώς ήρθατε. Την ε, κυρία Ίγκριντ Μασκάουζεν, μέλος της Αυστριακής Βουλής. Καλά τα λέω. Α, εκπρόσωπος της Eurojust μάλιστα. Και μάλιστα είστε εκπρόσωπο τη Αυστρία στη Eurojust. Ωραία. Τον κύριο Τζοβάνι Κέσλερ, Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ, τη Υπηρεσία Καταπολέμηση τη Απάτη ει βάρο των ε, κοινοτικών συμφερόντων. Και τον κύριο Χόλγκερ Ματ, Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ποινικολόγων. Καλώ ήρθατε. Η κυρία Καραμαλή έχει το λόγο. Merci, Monsieur le euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, συνάδελφοι βουλευτές. Πρώτα-πρώτα συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή των ε, Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης και ε, ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο, τον κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ, που οργανώσατε αυτήν την διακοινοβουλευτική εκδήλωση διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ευρωβουλευτές αλλά και οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων να προβαίνουν σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος της Στοχόλμη για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα, τα οποία ε, βεβαίως ε, μας οδηγούν στο ότι θα πρέπει να βιώσει προσοχή μας στην δικαστική αστυνομική συνεργασία, κάτι το οποίο ε, αφορά και τη συνθήκη της Λισαβόνας, διότι η συνθήκη αυτή ε, εθέσπισε ε, τον συνομοθέτη που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα και επίσης αναβαθμίστηκαν και τα εθνικά κοινοβούλια για τα θέματα τα νομοπαρασκευαστικά. Δεν θα μακρηγορήσω <clears throat> όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού ε, τον κανονισμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αμέσο μέλλον πρόκειται να κατεβάσει, πρόκειται να παρουσιάσει για την Eurojust γιατί έχουμε επομένω ε, τις πληροφορίες ε, που έχουν πει ότι έτσι πρόκειται να βελτιωθεί ε, η διεκπαιρέωση του διοικητικού έργου που τώρα είναι αρκετά χρονοβόρα. Πρόκειται για βήμα προόδου, έτσι πρόκειται να είναι πιο αποτελεσματική η Eurojust. Έτσι ε, οι εθνικές υπηρεσίες μπορούν να ε, επίσης λειτουργούν καλύτερα ε, και να επιχειρούν καλύτερα. Επίσης με τον νέο κανονισμό διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων για το έργο της Eurojust. Βέβαια, δεν προβλέπεται ε, να έχουμε ε, ποινικέ έρευνε όπω ορίζει το άρθρο 85 συνθήκη. Παρ' όλα αυτά όμω η ρύθμιση είναι λογική. Ε, ήταν δύσκολο να έχουμε παράλληλε διαπραγματεύσει. Πρώτον όσον αφορά τον εισαγγελία και από την άλλη μεριά όσον αφορά τι ποινικέ έρευνε από την Eurojust. Οπότε ε, σα τονίζω ότι η αναβάθμιση των ορμητήτων τη Eurojust αυτό είναι κάτι το απαραίτητο το οποίο συνοδεύει την θέσπιση του Ευρωπαίου Εισαγγελέως διότι ε, το πιο πιθανό είναι ότι ε, δεν θα καλύπτονται όλα τα κρατη Επίσης, ε, πριν έχουμε την αλλαγή της σημερινής ρύθμισης θα πρέπει να κάνουμε μία αξιολόγηση του πώς θα γίνει η μεταφορά αυτή τη απόφαση της 16 η 12 του 2008 που αφορά την Eurojust πώς θα μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο γιατί κάποια κράτη δεν έχουν μεταφέρει την απόφαση αυτή όπω η Γαλλία. Όμως σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να θεσπίσουμε ένα νόμο για να έχουμε την ενσωμάτωση τη απόφαση αυτή στο δίκαιό μα. Θα έχουμε επομένω αυτήν την ε, θέσπιση του, της του Ευρωπαίου Σαγγελία θα συνδέεται με Eurojust. Ε, για πρώτη φορά αυτή η ιδέα για τον Ευρωπαίο Σαγγελία ξεκίνησε από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Κλάους Χένς, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος και σε επίπεδο πανεπιστημιακό επίση το 1997 ε, αυτό υπήρξε ως ιδέα από κάποιους συμπληρώνομενες ο Ντελμάς Μαρτί, ως καθηγητής, πανεπιστημιακός και στην αρχή αυτό θεωρήθηκε ε, υπερβολικό αλλά τώρα αυτό ενσωματώθηκε στη συνθήκη ως μια δυνατότητα. Και αυτό από τότε που άρχισε να ισχύει με το άρθρο, ε, η συνήθεια Λισαβόνας και συγκεκριμένα στο άρθρο 86. Οπότε η Άνω και η στην ε, Γαλλία αναφανδώνεται υπέρ αυτής της ιδέας όπου είπαμε ότι θα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Επίσης το, η Εθνοσυνέλευσή μας ε, πέρασε δύο ψηφίσματα όσον αφορά αυτό τη θέση του Ευρωπαίου Αγγελέου πριν από 10 χρόνια. Ε, πάνω από 10 χρόνια, το 2002 και είχαμε τότε την πράσινη βίβλο της Επιτροπής για τον Εισαγγελέα. Ε, επίσης άλλο ψήφισμα το 2011 τον Αύγουστο με πρωτοβουλία δική μου. Και τότε είχαμε πλειοψηφία και σήμερα υπάρχει. Και επίσης σας τονίζω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ε, το οποίο συγκεντρώνει τη συνένεση από όλες τις πολιτικές πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Επίσης, η Εθνική Συνέλευση ε, ε, συνεργάστηκε με το Συμβούλιο Επικρατής του 2011 και επίσης και η Γερουσία το 2013 τον Ιανουάριο επίσης ψήφισε ένα κείμενο για το ίδιο αυτό ζήτημα. Ε, οπότε βλέπουμε ότι όλες οι πτέρυγες αυτές της πολιτικής μας ε, θέλουν να υπάρχει η Ευρωπαϊκή και έχουμε επίσης εργασίες, ε, ξερώνουμε με 10 κράτη-μέλη, έχουμε μια κοινή θέση και οι Υπουργοί Γαλλίας και Γερμανίας ε, συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 2013, γιατί είπαμε άμα έχουμε αυτή την ε, Ευρωπαϊκή, Εισαγγελία θα πρέπει να δούμε τις διαφορετικές ε, επιλογές και ενδεικτικά σας αναφέρω τι προτιμάμε αυτές τις δυνατές επιλογές. Το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να κρυφθεί είναι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Αγγελέα. Μπορούμε να πούμε ότι θα ασχοληθεί μόνο από τα οικονομικά σφαίρα της Ένωσης ή μπορούμε να πούμε ότι οι αρμοδιότητες αυτές θα αφορούν και ε, τα σοβαρά εγκλήματα. Αυτά που έχουν χαρακτηρία διασυνοριακό όπως ορίζει το 86 παράγραφος 4 της συνθήκης. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση επ' αυτού ξεκάθαρη είπε ότι η Ευρωπαϊκή Αγγελίας πρέπει να ασχολείται με το σοβαρό έγκλημα ε, όταν έχει δύο συνολικό χαρακτήρα. Ε, ε, επίσης για τη διακίνηση ανθρώπων, για την, ε, και το κυβερνό έγκλημα, για την τρομοκρατία, γιατί έχουμε το άρθρο 86 παραγραφό 4 της που ορίζει ότι ομόφωνα θα πρέπει να αποφασιστεί μια τέτοια παρέκταση αρμοδιοτήτων. Όμως αν έχουμε διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, κατά τη γνώμη μου, είναι δυνατόν να ισχύσει το άρθρο 330 της συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο μόνο τα κράτη τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία ε, θα ε, πρέπει να ψηφίσουν. Επομένως δεν προϋποτίθεται ε, η ομοφωνία ή φαστεί κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο, μια άλλη επιλογή είναι ο συλλογικός χαρακτήρας του Ευρωπαίου Εισαγγελία. Να έχουμε έναν και να έχει βοηθού από κάθε κράτο μέλος ή θα, υπάρχει, θα είναι συλλογικό όργανο, δεν θα είναι μόνο ένας ο Ε, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά το να είναι ένας. Γιατί θεωρεί ότι δεν θα είναι αποτελεσματική η εισαγγελία εάν έχουμε τέτοιο συλλογικό όργανο, ούτε οι έρευνε. Και ε, η Γαλλία όμω δεν συμφωνεί. Η Γαλλία θα προτιμούσε ένα συλλογικό όργανο, μια συλλογική εισαγγελία. Αυτό δεν θα παραβλάψει την ε, αποτελεσματικότητα. Έτσι θα υπάρχει άμεση σχέση με τα κράτη-μέλη και επομένως εάν η κάθε δικακή τάξη κράτους μέλους έχει αποδεχτεί το θεσμό θα είναι πιο αποτελεσματικός. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο καταστατικό, έτσι θα έχει περισσότερη νομιμοποίηση ο, ο εισαγγελέα. Αυτή η συλλογική φύση δεν θεωρούμε ότι θα στερήσει από την εισαγγελία την αποτελεσματικότητα. Θα υπάρχει βέβαια κάποιος πρόεδρος, κάποιος ε, ο οποίος είναι πρώτος μεταξύ ίσων με τους άλλους εισαγγελείς και αυτός θα μπορεί να ασκεί τις ε, διώξεις, θα μπορεί να, να πέμπει τις ε, υποθέσεις όποτε χρειάζεται και μπορεί να υπάρχει κυκλική αναλλαγή σε αυτή τη θέση. Και για κάθε υπόθεση που θα ορίζεται κάποιο εισηγητή από του εισαγγελεί που θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Σήμερα με το άρθρο 86 επίση προβλέπεται ε, να, να, να, να, να, να ξεκινάει από την Eurojust η οποία και εκείνη έχει συλλογική ε, φύση, συλλογική δομή. Τώρα, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά για τι ισχύει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα, ίσως από εκεί να προέρχονται ε, οι εισαγγελείς, αν βέβαια ε, έχουν τα σχετικά προσόντα και θα πρέπει να έχουν επίσης και την ανάλογη μακρά εμπειρία. Τέταρτο ζήτημα. Σε σχέση με το εφαρμοστείο δίκαιο. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει βέβαια κάποια δικονομία και το πιο ρελιστικό είναι να γίνεται όσο πιο συχνά παρα, παραπομπή και αναπομπή των υποθέσεων ε, σε εθνικές ε, εισαγγελίες και τώρα όσον αφορά τις ε, κυρώσεις και την άσκηση δίωξης θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει δυνατότητα να, να διαλέγει κανείς το που θα προσφύγει για να αποφύγει τις ε, πιο ε, αυστηρές κυρώσεις. Και αυτό προβλέπεται στο άρθρο 83 ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί και ένα τελευταίο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, να δούμε τι θα επιλέξουμε, είναι πώς θα ασκείται η εποπτεία επί της εισαγγελία. Θα πρέπει να μην υπάρχουν συγκρούσεις γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ένδικο μέσο ούτως ώστε να μπορεί κανείς να προσφύγει ε, σε δικαστήριο του κράτους ε, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση και έτσι να έχει τη δυνατότητα της ανατροπής μιας καταδίκης. Αυτά και είμαι στη διάθεση των μελών για ερωτήσεις τυχόν. Ευχαριστούμε κυρία Καραμαλή, λέει ο Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 12.30. Οπότε παρακαλώ ο καθένας να κάνει μια εισήγηση δεκαλέπτου για να έχουμε και χρόνο να συζητήσουμε με τους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές. Δεύτερος τώρα, θα λάβει το λόγο η κυρία Μάσουλ Κλάουζεν από τη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη γιατί στο πρόγραμμά σας αναφέρει πως θα ερχόταν ο αντιπρόεδρος της Eurojust, ο Κάρλος Ζέιεν. Δυστυχώς δεν ε, μπόρεσε να έρθει σήμερα, μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα 10 λεπτά, αν και πρέπει να παραδεχτώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί με τα θέματα που συζητάμε εύκολα θα μπορούσε να γεμίσει κανείς βιβλία. Όσον αφορά τώρα το πλαίσιο της ε, δικαστικής ε, συνεργασίας και τι μπορεί να βελτιωθεί έχουμε το ζήτημα της αμοιβιάς αναγνώρισης ε, η οποία είναι πραγματικά η βάση του χώρου δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Λισαβόνας και βέβαια πρέπει να ενισχυθούν τα δικονομικά δικαιώματα. Όλα αυτά βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των δικαστών και εισαγγελέων αμοιβαία και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο του νομικού πλαισίου και ακούσαμε μόλις τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι κοινέ ομάδες έρευνας όσον αφορά την αντιμετώπιση διασυνεργειακών οργανώσεων, εγκληματικών οργανώσεων. Αλλά οι κοινέ ομάδες έρευνας κοστίζουν. Γι' αυτό η χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας έχει μεγάλη σημασία. Η Eurojust ε, χρηματοδοτεί επιτυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια κοινές ομάδες έρευνας και έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των δικαστικών αρχών, των εισαγγελέων και των δικαστών. Έχουμε αποκτήσει μεγάλη πείρα στην σύσταση κοινών ομάδων έρευνας, το πώς να βοηθήσουμε στη σύστασή τους και το πώς να τις ε, χρηματοδοτούμε. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, ε, εγώ τώρα έχω κάποια αιτήματα από εσάς. Και εν ώψη των ε, εργασιών για την πρόταση ενός κανονισμού Eurojust θα σας αναπτύξω αυτά τα αιτήματα. Το πρώτο αίτημα είναι πώς η Eurojust θα ήθελε να αναγράφεται ρητός στο κείμενο του κανονισμού πως ένα από τα καθήκοντά της είναι η χρηματοδότηση των κοινών ομάδων έρευνας. Πρέπει να ευρεωθεί ο ρόλος της Eurojust. Συμφωνούμε όλοι πως αμοιβαία εμπιστοσύνη των δικαστικών αρχών, όπως αναφέρθηκε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να υπάρχει ένας αποτελεσματικός χώρος ποινική δικαιοσύνης. Επίσης θεωρούμε πως πρέπει να βελτιωθεί και η εκπαίδευση, οι ανταλλαγές, οι επισκέψεις, μελέτης και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Eurojust δηλαδή μαζί με τη Europol ε, μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την οικοδόμηση αυτής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ποια είναι τώρα τα ζητήματα προτεραιότητας κατά την άποψη της Eurojust που πρέπει να εξεταστούν ε, στην ε, επικείμενη πρόταση κανονισμού. Προφανώς το άρθρο 85 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί τον συντονισμό ως ε, τη βασική λειτουργία της Eurojust. Τι χρειάζεται η Eurojust λοιπόν για να επιτελέσει αυτό το ρόλο Πρώτα απ' όλα πληροφορίες. Πληροφορίες ε, για μία ποινική ε, εγκληματική δραστηριότητα και για μία έρευνα η οποία λαμβάνει η χώρα. Και αυτό είναι το δεύτερό μου αίτημα. Φροντίστε το κείμενο του κανονισμού να είναι τέτοιο ώστε να λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε την ε, λεγόμενη ευρωπαϊκή διάσταση, δηλαδή να μπορούμε να δρούμε προληπτικά και να μην αναμένουμε να απευθυνθούν σε εμάς οι δικαστικές αρχές με συγκεκριμένο αίτημα ε, αρρωγής, αλλά να μπορούμε προληπτικά και ε, με δική μας πρωτοβουλία να προσφέρουμε την βοήθειά μας για να αντιμετωπιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση ενός διασυνοριακού εγκλήματος. Αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το άρθρο 13 της απόφασης περί Eurojust, αλλά δεν το έχουν εφαρμόσει όλα τα κράτη-μέλη, εφαρμογή καθυστερή και αυτό φαίνεται και από την ε, έκτη αμοιβαία αξιολόγηση που λαμβάνει η χώρα. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τη Europol, να λαμβάνουμε πληροφορίες από τη Europol Προφανώς το ίδιο ισχύει και για τον Όλαφ, την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης. Θα επανέλθω στο πρώτο μου αίτημα, τις κοινέ ομάδες έρευνας και την χρηματοδότησή τους. Το ζήτημα των περαιτέρω αρμοδιοτήτων ε, προφανώς είναι ένα επίμαχο ζήτημα η κατάσταση έχει ως εξής. Οι αρμοδιότητες των εθνικών μελών διαφέρουν και προφανώς αυτή η κατάσταση δεν είναι ιδεώδης. Μάλιστα έχουμε συναντήσει περιπτώσεις όπου είχαμε προβλήματα λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στις αρμοδιότητες των εθνικών μελών. Όμως προφανώς επαφίεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους πολιτικούς να κρίνουν εάν θα πρέπει να έχει περαιτέρω αρμοδιότητε η Eurojust όπω η πιθανή έναρξη ερευνών ή η διερεύνηση τυχών ε, συγκρουόμενων δικαιοδοσιών μέσω της έκδοσης μια δεσμευτική απόφασης. Εάν κρίνεται πως θα πρέπει να αποκτήσει περαιτέρω αρμοδιότητες η Eurojust, πρέπει να εξετάσουμε ορισμένα πράγματα όπως ε, παραδείγματος ε, χάρη η δυνατότητα προσφυγής ε, εναντί αυτών των αποφάσεων, τα ουσιαστικά κριτήρια για δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, η συνέχεια η οποία δίνεται σε μια απόφαση για την έναρξη μιας έρευνας και πρέπει επίσης να δούμε και τον αντίκτυπο αυτών των αποφάσεων στην αρχή της ε, νομιμότητας, ε, ενώ εδώ πέρα δηλαδή την ε, υποχρεωτική δίωξη. Κάποια ζητήματα λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε. Επίσης γνωρίζουμε πώς θα προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν την κοινοβουλευτική εποπτεία της Eurojust, κάτι το οποίο ορίζουμε, την εμπλοκή δηλαδή του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων στις ε, δραστηριότητες της Eurojust. Θεωρούμε πως η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ενισχύσει την δημοκρατική λογοδοσία της ε, Eurojust και θα ενισχύσει και την σχέση μεταξύ Eurojust και Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα, τι πρέπει να αξιολογηθεί. Θεωρούμε πως η αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάσει την ικανότητα της Eurojust να κληρώσει την αποστολή της ε, και τους στόχους της, ειδικά το εάν ε, συμφέρει οικονομικά η λειτουργία της Eurojust. Θεωρούμε πως η ανεξαρτησία της Eurojust όσον αφορά τις ε, μεμονωμένες περιπτώσεις ε, το επιχρησιακό σκέλος πρέπει να διατηρηθεί. Γι' αυτό η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να κρίνει ε, συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ποινικού δικαίου. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση. Όπως είπε και η Επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ, αυτό είναι δικό σας θέμα, εσείς θα το οργανώσετε, εμείς δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη άποψη, αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μας είναι να υπάρχει μία αξιολόγηση από όλα τα θεσμικά όργανα και τους φορείς και να μην καταλήγουμε να κάνουμε πολλές φορές τα ίδια πράγματα ή, ακόμη χειρότερο, με αντιφατικά αποτελέσματα. Δεν θα το θέλαμε αυτό. Γι' αυτό κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρχει μία κοινή αξιολόγηση. Μία κουβέντα ακόμα για, τον, ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και η κυρία Καραμαλή, εμείς θεωρούμε πως ε, προφανώς ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Eurojust πρέπει να συνεργάζονται στενά πρέπει να υπάρχει αμοιβαία στήριξη, συμπληρωματικότητα και συνέργειες και προφανώς εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συσταθεί ε, όχι μόνο ε, αν, στη, όχι με τη συμμετοχή όλων των κρατών θα πρέπει να υπάρχει προφανώ και μια συνεργασία με τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα συμμετέχουν, αλλά και με τρίτες χώρες. Και τέλος αναφέρθηκε πως το άρθρο 86 αναφέρει πως ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να προκύψει μέσα από την Eurojust. Πράγματι μπορεί να αντλήσει τους ε, πόρους που έχει στη διάθεσή της η Eurojust και ε, θα μπορούσαν ακόμα και να συστεγαστούν οι δύο υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας από τη Eurojust και πάμε τώρα ε, στην παρουσίαση του εκπροσώπου της Όλαφ, του κ. Τζοβάνι Κέσλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές και ευρωβουλευτές, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για την συνεχιζόμενη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την δημιουργία του γραφείου εισαγγελίας. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και η Γενική Διεύθυνση Όλαφ κάνουν αυτό το συντακτικό έργο από πλευράς Κομισιόν. Φυσικά ε, την πολιτική ευθύνη έχει ε, η Επίτροπος Μάλστρομ και ο Επίτροπος Εμέτας. Η δουλειά της Κομισιόν έχει φτάσει σε, προχωρημένη, σε προχωρημένο στάδιο και πρέπει απλώς το Σώμα των Επιτρόπων να εγκρίνει το τελικό κείμενο, κάτι που θα γίνει σε επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Ποτέ δεν ξέρει κανείς μέχρι να συμβεί κάτι πότε ακριβώς θα εγκριθεί στην Κομισιόν. Α πούμε, ας πούμε για να είμαστε σίγουροι, φέτος ότι θα γίνει. Αρκετά σύντομα δηλαδή. να σας πω μερικές σκέψεις για αυτό το θέμα από πλευράς μας. Καταρχάς, πρέπει να καταλάβουμε πού ξεκινάμε. Ποιες είναι οι υποθέσεις μας. Δεν, κάνουμε, δεν φτιάχνουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο και μόνο για το λέει συνθήκη. Υπάρχει πολλή δουλειά που έχει γίνει στην αρχή. Θα τα πω λίγο μα, γιατί προσπαθώ να είμαι σύντομος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σημερινό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας όλοι είναι να αντιμετωπίσουμε το διεθνές, διασυνοριακό δηλαδή έγκλημα και μάλιστα διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα. Και το πλαίσιο που έχουμε για να το αντιμετωπίσουμε είναι ανεπαρκές. Είναι το σύστημα του 19ου αιώνα που βασίζεται στην εθνική άποψη, ας πούμε, εθνική προοπτική και εθνική θεώρηση. Κάθε χώρα ασχολείται με τις δικές της υποθέσεις, τα πλαίσια των δικών εθνικών αρμοδιοτήτων, βασιζόμενες στις δικές εθνικές υπηρεσίες. Λες και, λες και υπάρχουν ακόμα εθνικά εγκλήματα και μόνο. Υπήρχαν ίσως το 19ο αιώνα, αλλά όχι πια. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά από την δική μας εμπειρία στην Όλαφ. Αυτά τα εγκλήματα, όλο και περισσότερο, αν όχι πάντα, έχουν διασυνοριακή φύση. Αλλά εμείς τα αντιμετωπίζουμε σαν τα εθνικά. Δηλαδή με τελείω κατακαιρματισμένο τρόπο. Οι υπηρεσίε που έχουμε, οι ερευνητικέ, οι εθνικές δικαστικές και εισαγγελικέ υπηρεσίε, ασχολούνται Αντιμετωπίζουν όμως κυρίως διασυνοριακά, διεθνικά φαινόμενα, αλλά με εθνική προοπτική. Άρα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα και συνολικά το έγκλημα. Τέλο πάντων, και όταν το βλέπουμε, βλέπουμε ένα κομμάτι του. Και αν είμαστε τυχεροί, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία και άλλες πληροφορίες σε άλλες χώρες. Και έχουμε λοιπόν το σύστημα μετά της διεθνούς συνεργασίας. Καλό είναι αυτό, αλλά πάντα ξεκινάμε από την διεθνή, συγγνώμη, από την εθνική σκοπιά και μετά πάμε στη διεθνή συνεργασία, η οποία ακόμα και σήμερα βασίζεται στο μοντέλο του 19ου αιώνα, στην, α, της αμοιβαίας δηλαδή δικαστικής συνδρομής. Αυτό δεν αρκεί. Ο Ευρωπαίος εισαγγελέα λοιπόν θα είναι το επόμενο βήμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα είναι το επόμενο βήμα και θα αντιμετωπίζει τα εγκλήματα αυτά όχι από εθνική σκοπιά αλλά από ευρωπαϊκή σκοπιά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ευρωπαϊκά φαινόμενα από τη γωνιά σου, στο γραφείο σου, στη χώρα σου. Αυτή λοιπόν αυτό είναι το όραμα. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα έχουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο εισαγγελία. Γραφείο. Κυρία Καραμαλή, ξέρουμε ήδη να λειτουργούμε με συλλογικό τρόπο. Τη θέση σας ε, θα τη συζητήσουμε ε, στο Συμβούλιο όταν παρουσιαστεί. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα τη συζητήσουν και τα εθνικά κοινοβούλια προφανώς και το ευρωπαϊκό συνεχεία. Αλλά όμως δεν υπάρχει κανένα δικαστικό γραφείο ή εισαγγελικό γραφείο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα που να βασίζεται σε αυτό το συλλογικό μοντέλο. Δηλαδή κανένα εθνικό γραφείο εισαγγελία δεν είναι συλλογικό, δεν είναι ευρωπαϊκό. Ε, η συλλογική μορφή είναι καλή γιατί ενισχύει και προσαυξάνει τη διεθνή συνεργασία. Πιστεύουμε ότι το αμυγός συλλογικό μοντέλο είναι ασύμβατο με την έννοια του γραφείου. Γραφείο. Δεύτερο, το συλλογικό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά για τη Eurojust. Γιατί, δηλαδή για τη διεθνή συνεργασία, δεν είναι πάλι συμβατό με την έννοια της ανεξαρτησίας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας σε αντιδιαστολή με τη Eurojust δεν θα απαρτίζεται αυτό το σώμα από διορισμένους εισαγγελείς από τα κράτη-μέλη. Θα είναι ένα σώμα ανεξάρτητο. Εν πάση περιπτώσει, είπατε δεν είναι. Τι είναι το μοντέλο μας. Δεν είναι ένα χταπόδι το οποίο θα βρίσκεται ας πούμε στις Βρυξέλλες με πλοκάμια σε όλα τα κράτη-μέλη. Όχι. Δεν είναι χταπόδι. Θα είναι ένα αποκεντρωμένο μοντέλο όπως το λέμε, ή ενοποιημένο αν προτιμάτε μοντέλο, δηλαδή ένα γραφείο που θα αποτελείται από εισαγγελείς, που θα έχει ένα μικρό κεντρικό γραφείο, συντονιστικές αρμοδιότητες και θα απαρτίζεται από εισαγγελείς κρατών μελών που θα τους βρούμε στα κράτη-μέλη, θα είναι εισαγγελείς από τα κράτη-μέλη, και θα κάνουν τη δουλειά, θα συνεχίζουν τη δουλειά των κρατών μελών. Δηλαδή, ε, ενοποιούμε την Εθνική Εισαγγελία, τις Εθνικές μάλλον Εισαγγελίες, ε, και τις φέρνουμε σε επαφή με άλλες Εθνικές Εισαγγελίες, χάρη σε αυτό το κεντρικό γραφείο που θα έχει συντονιστικό ρόλο στις Βρυξέλλες, περίπτωση αν εδρεύει στις Βρυξέλλες. Αυτό το κεντρικό γραφείο θα έχει την ευρωπαϊκή θεώρηση. Τι άλλο πλεονέκτημα θα έχει. Θα εφαρμόσει για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης. Αυτή την φοβερά σημαντική έννοια ε, που προκύπτει από την Στοχόλμη, το πρόγραμμα της Στοχόλμης, πουθενά δεν τη βλέπουμε υλοποιημένη. Για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δημιουργήσουμε τελικά αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελίας, θα ξεπεράσουμε το θέμα της αμοιβαία νομικής ή δικαστικής συνδρομής. Σήμερα, αν ένας εισαγγελέας από τη Βόρεια Ιταλία, όπως ήμουν εγώ, ε, ήθελε να πάρει αποδεικτικά στοιχεία από την Αυστρία, ας πούμε, πέρα από τα σύνορα, ας πούμε, θα έπρεπε να κάνει ολόκληρα διαβήματα. Αύριο με το γραφείο αυτό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα έχουμε Ιταλούς, Γερμανούς, Αυστριακούς, Γάλλους εισαγγελείς που θα ανήκουν στο ίδιο γραφείο, στο ΕΠΟ αυτό όπως το λέμε, το ακρονιμιό του είναι. Επομένως η συνεργασία μεταξύ του δεν θα είναι πλέον διεθνή συνεργασία, θα είναι συνεργασία μεταξύ μελών του ίδιου γραφείου. θα ξεπεράσουμε την ανάγκη για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή. Με τρομερά ωφέλη θα αποφεύγουμε φυσικά και τη σπατάλη του χρόνου και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Καιρός να κλείσω όμως. Για το θέμα της αρμοδιότητας, δύο λόγια. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσει με αρμοδιότητες ε, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους ομοφωνίας, για να μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση. Και για να συμμετάσχουν τον περισσότερες χώρες σε αυτό το γραφείο Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Βεβαίως αυτό το γραφείο σκοπεύουμε να το επανδρώσουμε ε, βασιζόμενοι στους πόρους που έχουμε ήδη. Και επίσης θα στηθεί με κόστος μηδέν εντό αγωγικών, εν Θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς που έχουμε. Θα είναι ένα γραφείο που θα βασίζεται στους ανθρώπινους ε, και οικονομικούς πόρους ε, που έχει η ΟΛΑΦ, η Eurojust και τα Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Δέκα λεφτά Dan, κάνατε. Και τώρα έχουμε τον κύριο Χόλγκερ Ματ που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποινικολόγων θέτουμε το πλαίσιο για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το νέο μόρφωμα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελίας. Έτσι λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίζει το ρόλο της, ούτως ώστε να διώκονται και να δικάζονται ε, υπεύθυνοι για σοβαρά διασυνοριακά εγκλήματα. όπως προβλέπει με βάση τη διατάξεις δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ποινικού δικαίου. Κύριε Ματ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κοίταξε, αυτέ τι προτάσει δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί οριστικά. Οπότε τι να κάνω, και εγώ θα, ε, προσπαθήσω να σα πω όσο μπορώ καλύτερα αυτά τα οποία σκέφτομαι. Βέβαια ο κύριο ε, Τζοβάνι εδώ, <laughs> παρακαθήμενος, Βεβαίω από την όλα πρόκειται τα ξέρει καλύτερα από μένα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, τη, με την Ευρωπαία Εισαγγελέα με αυτή την καινούργια υπηρεσία. Πρώτα-πρώτα. Θα σας πω ότι εκπροσωπώ την Ένωση Ευρωπαίων Ποινικολόγων και καλύπτουμε 35 με 40 χώρες. Την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και χώρες εκτός αυτής. Παρακολουθούμε όλες τις προτάσεις που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχολιάζουμε, συμμετέχουμε σε συναντήσεις ε, των ειδικών, οπότε δεν μπορώ παρά να σταθώ στην ιστορική ψηφοφορία της ε, Επιτροπής όσον αφορά την οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Δυστυχώς βέβαια δεν εγκρίθηκαν, δεν καλύφθηκαν όλες μας οι προτάσεις. Παρ' όλα αυτά. Θεωρούμε πολύ θετική αυτή την ψηφοφορία. Ήταν ένα ιστορικό βήμα σε σχέση με αυτόν τον χάρτη πορείας που είναι τμήμα του προγράμματος της ε, Στοκχόλμης. Οπότε για αυτόν τον τρόπο βοηθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστούμε βέβαια και την κυρία Αντωνέσκο που ήταν η εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Αντωνέσκο επέδειξε αφοσίωση στο έργο της, διπλωματικές ικανότητες και κατανόηση των θεμάτων κατά προγραμματεύση. Οι βασικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τον Ευρωπαίο Αγγελία, ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί οριστικά. Προβλέπεται ένα συγκεντρωμένο σύστημα, προβλέπεται ευρωπαϊκή συνεργασία με την Europol, την Eurojust, με την Olaf, προβλέπεται να υπάρξει ανεξαρτησία του θεσμού αυτού, να διέπεται από δημοκρατικό έλεγχο και υποχρέωση λογοδοσία, δικαστικό έλεγχο, να υπάρχει κάποιο δικονομικό πλαίσιο στο οποίο να κινείται και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επίση, ασκεί ποινικέ διώξει, έρευνε. Και επομένως με δεδομένα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης Έχουμε επισημάνει 14 σημεία στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Δεκατέσσερα σημεία λέγω στα οποία στάθηκε η Ένωση Ευρωπαίων Ποινικολόγων. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τον φορέα των διοικητικών συλλόγων πολλών χωρών και με γερμανικούς νομικούς φορείς επίσης. Να σας παρουσιάσω αυτά τα 14 σημεία που έχουν κυρίως πολιτικό χαρακτήρα. Πρώτα πρώτα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ε, ενδείξεις. Κύριε Κέσλερ, καταλαβαίνω ότι και εσείς χρειάζεται το να έχετε, ε, να έχετε κάποιες ενδείξεις ότι πρέπει να υπάρχει αυτό, αυτή, αυτή η υπηρεσία. Οπότε θέλω επομένω και εσείς να το, να το συμμεριστείτε αυτό, να συμφωνήσετε. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός ότι να χειρίζεται ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας τις υποθέσεις που δεν χειρίζονται τα κράτη-μέλη. Άρα να υπάρχει κάποιο είδους συμπληρωματικότητα. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει και η αναλογικότητα. Και αυτό το ορίζει το άρθρο 86 της συνθήκης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ίσο, ίση μεταχείριση, ίσες δυνατότητες ε, μεταξύ εθνικών εισαγγελιών και του Ευρωπαίου εισαγγελία. Αυτό να ισχύσει και για την νομική αρρωγή γιατί βέβαια εδώ πέρα βλέπουμε ότι θα χρειαστούν παραπάνω πόροι, αλλά αν θέλουμε να έχουμε ουσιαστική προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει και με αυτή τη νέα υπηρεσία κάτι τέτοιο να γίνει όσον αφορά την, ε, την του έργου της. Να υπάρχουν επίσης κάποιες ευχαριστικές ε, δικλίδες. Και στην ΦΕΑ περιοχή πριν τη διεξαγωγή της έρευνας να λάβουμε επίσης υπόψη την οδηγία για τα ελάχιστα πρότυπα. Κατά αυτόν τον τρόπο να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη προς αυτό το νέο θεσμό. Τώρα η συλλογή των αποδείξεων. Και αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί και επίση πάλι στην ε, ασαφή περιοχή ε, πριν την ε, δύναμη μια Να δούμε επίση να μην έχουμε form shopping, δηλαδή την, την, δυνατότητα αναζήτηση τη πιο βολικής ενόμης και να υπάρχουν και οι εγγύησει σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Υπάρχει βέβαια δικαστικό έλεγχος επί αυτή τη ε, υπηρεσία. Και να αφορά κάθε απόφαση, ακόμα και αρνητική απόφαση. Έβδομο σημείο. Να ρυθμιστούν οι αρμοδιότητες αυτής της υπηρεσίας, αλλά και της Eurojust και της Olaf και της Europol σε σχέση με αυτή την υπηρεσία. Όγδον, πολιτικός δημοκρατικός έλεγχος. Ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα και υποχρεώσει λογοδοσίας. Συντονισμός με τις εθνικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο προβλέπεται, αλλά στην πράξη ε, για τα ποινικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να δούμε, προς ενδιαφέρον, τι λύση θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού. Δέκατον. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Non bis in idem. Επίσης, τι θα γίνει στις ε, μικτές υποθέσεις σε αυτή την περίπτωση ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα ασχολείται με αυτές τις μικτές υποθέσεις και που αφορούν επίσης τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Τέλος, κανόνες για την άσκηση ποινική διώξεως, παραπομπή σε δίκη και επίσης για τα 11 μέσα, Ούτως ώστε πάλι να δούμε πώς δεν θα μπορεί κάποιος να επιλέξει το πιο βολικό δικαστήριο σαν διάδικος. Επίσης, μηχανισμοί αποζημίωσης σε περίπτωση που έχουμε καταχρηστική άσκηση των καθηκόντων αυτής της ε, υπηρεσίας. Επίσης, να έχουμε υπηρεσίες διερμηνίας αλλά και μετάφρασης. να μην ξεχνούμε πάντως το ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρύθμιση ή κάποια δικονομία νομικά δεσμευτική να ισχύσει ό,τι προβλέπει το άρθρο 86 παράγραφος 3 της συνθήκης. Οπότε και αυτές οι δικονομικές διατάξεις να έχουν και τις συνήθεις δικονομικές ε, εγγυήσεις, αναγνώρισμα, αλλά επίσης να προβλέπεται και νομική αρρωγή κατά τη διαδικασία ενώπιον ε, του Ευρωπαίου Ισαγγελέα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι ε, έτσι λειτουργεί και το Κοινοβούλιο. Έχουμε τη διερμηνία, αλλά προβλέπεται μέχρι συγκεκριμένη ώρα. Προβλέπετε να έχουμε τους διερμηνείς μαζί μας μέχρι τις 12.30. Οπότε παρακαλώ, παρακαλώ θερμότατα, προσπαθήστε πολύ, πολύ, ούτω ώστε να, να, να κάνετε μονόλεπτες ε, παρεμβάσεις, άντε 1,5 λεπτό. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε δεύτερο γύρο παρεμβάσεων από το πάνελ. Για τις 12.30 περίπου θα φύγουν οι διερμηνείς. Θα έχουμε μόνο αγγλικά. Mr. Albrecht from the European Parliament. Thank you very much, Try to make it in one minute, please. And I will try to keep it. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, όσον αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το βασικό θέμα εδώ πέρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η εμπιστοσύνη των ε, κρατών μελών, ε, των αρχών, των εισαγγελέων και βεβαίω των πολιτών και του Κοινοβουλίου. Και δεν πρέπει νομίζω να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Όλαφ. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα παρόμοιο με τις ε, Eurojust, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 της συνθήκης, να υπάρχουν κοινές ε, οικονομικές ε, διαδικασίες ε, ανάλογες με των κρατών μελών και πάρα πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι εδώ και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα, το, ε, δεν θα ακολουθεί η γρήγορη διαδικασία, δεν πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα πλήξει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία των κρατών μελών. Αυτή η δήλωσή μου νομίζω ότι είμαι σαφής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μίκελσεν από την Ορβηγία. Η κυρία Μίκελσεν βεβαίως. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας φιλοξενεί σήμερα και προσκάλεσε και Νορβηγούς βουλευτές θίγονται κάποια επίκαιρα ζητήματα. Η δικαστική συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ατιμορρησίας σοβαρών εγκλημάτων. Βλέπουμε καμία φορά πως ε, εγκληματίες που κατηγορούνται για δολοφονία ή σεξουαλικά εγκλήματα φεύγουν από την χώρα όπου διαλύμα και πάνε στην ε, χώρα προέλευσής τους. Οπότε εδώ πέρα βοηθάνε πάρα πολύ οι συμφωνίες έκδοσης, αν και δεν αποτελούν εγγύηση βεβαίως, το καθιστούν πάρα πολύ ευκολότερο το να λογοδοτήσουν οι κατηγορούμενοι. Όμως συχνά οι πιθανοί δράστες πηγαίνουν σε χώρα τους η οποία μπορεί να μην έχει υπογράψει συμφωνία έκδοσης. Και έτσι έχουμε ατιμωρησία. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 2008 ένας ε, Νορβηγός φοιτητής ε, βιάστηκε και δολοφονήθηκε στο Λονδίνο. Η Βρετανική αστυνομία ε, εξέδωσε διεθνές ένταλμα για έναν υπήκο Ιεμένης ο οποίος κατέφυγε στη χώρα του αλλά δεν υπάρχει συμφωνία έκδοσης Βρετανίας Ιεμένης και κάθε προσπάθεια έκδοσης απέτυχε ζει ελεύθερος, τον προστατεύουν οι αρχές της χώρας, τους, της χώρας του και ε, προτάθηκε πως οι χώρες θα έπρεπε να μελετήσουν τη δυνατότητα σύστασης ε, μιας ε, ανεξάρτητης διεθνούς ε, νομικής αρχής για να μην υπάρχει ατιμορρησία σε τέτοιες διεθνείς ε, περιπτώσεις. Επιπλέον έχει προταθεί πως θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είμαι πεπισμένη πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διεθνείς ποινικέ περιπτώσεις και το ζήτημα της ατιμορρησίας. Επίσης, το έχω θέσει αυτό και στις συναντήσεις του ΟΑΣΕ άλλων διεθνών οργανισμών και ελπίζω στη μελλοντική μας συζήτηση να δούμε το πώς μπορούν να συνεργαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες ε, για να δούμε τι θα κάνουμε στις περίπλοκες ε, ποινικέ ε, υποθέσεις που εμπλέκουν τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Τάσκολα από την Ιταλία. Προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος έχω αμηχανίες, όχι πολιτικής φύσεως, αλλά νομικής φύσεως, για το, την προσωπικότητα αυτή του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Να σας πω ότι θα είναι πρώτη φορά που ένα γραφείο εισαγγελία θα λειτουργεί υπό τελείως διαφορετικές και ανομοιογενείς δικαιοδοσίες. Επομένως θα πρέπει να θέσουμε με πολύ σοβαρό τρόπο τον τρόπο που θα ασκεί την ποινική του δράση ο εισαγγελέα καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει. Όταν μιλάω για τρόπους άσκησης των δραστηριοτήτων στον ποινικό τομέα. Δεν, θα ξέρουμε, δεν ξέρουμε μάλλον ακόμα αν ο Ευρωπαίος Αγγελέας θα ασκεί αυτή την ποινική δράση με αποκλειστικό τρόπο ή παράλληλα με την Εθνική Εισαγγελία της αρμόδιας χώρας. αυτή την περίπτωση, στην δεύτερη περίπτωση τα δικαστικά προβλήματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Γιατί ο Ευρωπαίο αγγελία απλώ θα έπαιζε το συντονιστικό ρόλο, α πούμε, στο έργο των υπολείπων εισαγγελιών. Αν όχι, αν είχε αποκλειστική αρμοδιότητα, θα είχαμε τρομακτικά ε, νομικά προβλήματα. Και επομένω θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή του ουσιαστικού δικαίου, αλλά και του δικονομικού δικαίου που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Όλα αυτά τα προβλήματα επιλογής της δικαιοδοσίας που καθορίζονται από το είδος του εγκλήματος και θα επαυξάνονταν λόγω των προβλημάτων αρμοδιότητας που θα έχει ο καθένας ε, και σε ποια επικράτεια. Μιλάμε τώρα πάντα για διεθνές έγκλημα αυτά τα αδικήματα μπορεί να γίνουν σε διαφορετικές επικράτειες, όχι σε μία. Επομένως θα πρέπει να επιλέξουμε ποιο εθνικό ουσιαστικό δίκαιο ισχύει με βάση κάποια κριτήρια. Θα μπορούσε να είναι ο τόπος που διαπράχθηκε το έγκλημα, θα μπορούσε να είναι ε, το δίκαιο της χώρας που διαμένει ο κατηγορούμενος ή το θύμα. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και να δούμε πώς θα κάνουμε τις επιλογές μας. Ακούσαμε πολύ περίπλοκα σενάρια. Γιατί υπάρχουν προβλήματα σύγκρουσης δικαιοδοσιών και σύγκρουσης αρμοδιοτήτων όταν έχουμε πρόβλημα να εντοπίσουμε το, την επικράτεια που διαπράχθηκε το έγκλημα. Ή όταν διαπράχθηκε σε περισσότερες από μία επικράτειες. Ε, θα μπορούσε επομένως ο Ευρωπαϊκός Αγγελέας να δρά με βάση έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Ποινικού Δικαίου να ασχολείται με την προδικαστική έρευνα και να σταματάει εκεί η δράση του. Σε αυτή την περίπτωση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προδικαστικών ε, Ερευνών θα πρέπει να συντονιστεί με τα εθνικά συστήματα. Και θα είναι δύσκολος αυτός ο συντονισμός, γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα εγγύσεων που προβλέπονται στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Και σε ό,τι αφορά την Ιταλία, θέλω να σας πω ότι όχι μόνο ε, έχουμε πολύ περίπλοκες εγγύησεις που προβλέπουμε στη δικαιο... στην νομοθεσία μας. Έχουμε όμως και ένα άρθρο, το άρθρο 111 στο Σύνταγμα, που προσδιορίζει τα όρια των ερευνών ανάλογα με το ήθος του ε, αδικήματος. Να σας το πρόβλημα το χρονικό που έχουμε. Αμέσω μετά θα πάμε για το γεύμα. Αλλά έχω να σα υπενθυμίσω ότι μέχρι τι 12.30 έχουμε διερμηνία. Ο κύριο Φαν Κόστεν από την Ολλανδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ δε τα μέλη του πάνελ για την παρουσίαση που έκαναν. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς θα αποφύγουμε το ότι, γιατί το έχουν θίξει πολλές φορές συνάδελφοι στην συνάδελφη, να ε, απασχολείται ο Ευρωπαίος Εισαγγελίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ζητήματα τα οποία θα είναι πολύ περισσότερα και ευρύτερα από αυτά τα οποία αρχικά, για τα οποία αρχικά είχε προβλεφθεί. Σας ευχαριστώ κύριο Σκέλης από την Πολωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, αλλά το βασικό ερώτημα είναι το εξής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορέσει να εγγυηθεί την ε, νομική προστασία ή θα έχει την, ε, το προνόμιο του να ξεκινά με δική της ε, πρωτοβουλία έρευνες. Εγώ γνωρίζω το πολωνικό σύστημα και το πώς λειτουργεί εκεί η εισαγγελία και νομίζω πως θα πρέπει να δούμε το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή η αστυνομία συλλέγει τα στοιχεία και μετά είναι απόφαση του εισαγγελέα ή έρευνα ή όχι. Με την αύξηση λοιπόν των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περνάμε κατευθείαν στην έρευνα και θα είναι η μόνη προσέγγιση που υπάρχει. Σας ευχαριστώ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστώ εξ της Επιτροπής της Βουλής των Λόρδων για την ε, δικαιοσύνη, τα θεσμικά όργανα και την προστασία των ελπίζω να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διατήρηση του Eurojust ε, ανεξαρτήτως του opt-out που έχουμε για το άρθρο 36. Η συμμετοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ε, προστασία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε εποπτεία που θα ασκηθεί θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν μόνα τους τα κοινοβούλια και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να φτάνει όμως μέχρι του σημείου της, ε, των πληροφοριών για επιχειρησιακά ζητήματα. Θα πρέπει να βασιστεί η εποπτεία σε υφιστάμενους μηχανισμούς. Είμαστε υπέρ των κοινών ομάδων έρευνας και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα η Επιτροπή μου δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί αλλά η κυβέρνηση της χώρας μας είναι εναντίον και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει δημοψήφισμα. Σας ευχαριστώ και ο από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε με τις εισηγήσεις του Προεδρείου. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία, η θέσπιση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι μια πολύ σημαντική όθηση προς την ενίσχυση της ε, ε, δικαιοσύνη στον νέο ευρωπαϊκό χώρο. Το αν θα είναι ένα ή θα είναι εκ αυτό μικρή σημασία έχει. Μεγάλη σημασία έχει όμως πώς θα στελεχωθεί το συγκεκριμένο γραφείο από εθνικούς εισαγγελείς, οι οποίοι θα, θα συντονίζονται άμεσα με τον Εθνικό Εισαγγελέα, τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και έτσι θα αποφεύγουμε περιττή γραφειοκρατία και διαδικασίε γραφειοκρατικές που ξέρουμε πόσο πολύ κοστίζουν και σε χρόνο και σε χρήμα. Και τέλο, έναν κατάλογο κοινό μπορούμε να συμφωνήσουμε, πρέπει να συμφωνηθεί για τα εγκλήματα κατά του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κοινοτικών κοντιλίων, για τη λαφρομετανάστευση, τους διακινητές, του σύγχρονους δουλέμπορους, το εμπόριο λευκής σαρκός. Πιστεύω ότι ένας μικρός κατάλογος σαν πρώτη αρχή μπορεί να αποτελέσει προϊόν συνένεση και συμφωνίας όλων μας έτσι ώστε να κάνουμε το πρώτο και σημαντικό βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Συμπάνω πως βεβαίως ε, πράγματι για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ε, υπάρχει πρόβλεψη ποινικού δικαίου και έχουμε μία πρόταση ε, με μία σειρά ορισμών ακριβώς για τα ποινικά αδικήματα τα οποία θα συμπεριληφθούν και τις κυρώσεις που θα καθοριστούν ως ε, ελάχιστες ε, ε, προδιαγραφές για όλα τα κρατη Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Σέξμπορκ από την Γερμανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εθνικούς ε, βουλευτές ε, και ήρθαμε από μακριά, καλό θα είναι να έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε με διερμηνία. Όταν μιλάμε για τη συνεργασία νομίζω πως έχει αποφασιστική σημασία η συμπερίληψη των εθνικών ε, κοινοβουλίων Βεβαίω το άρθρο 86 μιλάει για αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε πάρα πολλά σημεία τίθεται ζήτημα επικουρικότητα. Ε, ε, οπωσδήποτε η, Βρετανική, η Γερμανική Βουλή, με συγχωρείτε, δεν είναι εναντίον, αλλά ε, βλέπει το θέμα και το εξτάζει με τρόπο κριτικό. Τίθενται πράγματι ζητήματα διαδικαστικά, αυτά τα οποία θα εξετάσουμε ιδιαίτερα όσον αφορά το εάν τηρείται η επικουρικότητα σε ζητήματα ποινική δικονομίας Βλέπω λοιπόν πως σε πάρα πολλά σημεία έχουμε προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, ζητήματα οργάνωσης, ε, νομιμοποίησης μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία ε, που θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετική από την Εθνική Εισαγγελία, πολλά λεπτομερή προβλήματα, παραδείγματο χάρη τι δικαίω, τι, ποιο δίκαιο θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στους υπόπτους, ε, ποια θα είναι η συνεργασία και πώς θα διασφαλιστεί η συνεργασία αυτής της υπηρεσίας με τις εθνικές αστυνομίες θα πρέπει να είναι πραγματικά άμεση και χωρίς ε, προβλήματα. Δύο ακόμα θέματα και τελειώνω, γιατί δεν το βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, περίπλοκες υποθέσεις, πώς θα ερευνηθούν από τις εθνικές αγγελίες, θα γίνει από τις εθνικές αγγελίες ή από την κεντρική υπηρεσία τι θα γίνει με παρακολουθήσεις ε, τηλεφώνων. Έχουμε αναλύσει το εθνικό δίκαιο. Ποιες είναι οι εγγύησεις που υπάρχουν. Ε, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια ζητήματα δικονομικά από πλευράς ε, Γερμανίας και δεν ξέρω, έρχονται και οι διακοπές, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε την προθεσμία των 8 εβδομάδων ε, πρέπει να το λάβει υπόψη της αυτό η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ που συνοψίσατε τις ανησυχίες σας. Το ίδιο ισχύει και για τους ομιλητές μας. Καταλαβαίνω πως έγιναν συγκεκριμένες ερωτήσεις προς δύο συγκεκριμένα μέλη. Ε, εκπρόσωπο της Eurojust θέλετε, θέλετε κι εσείς να αφαιρθείτε σε κάποια πράγματα βεβαίως. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μας βοηθήσετε γιατί προφανώς... Ε, οι διερμηνείς ε, ξεπερνάνε το ωράριό τους ε, και τους ευχαριστούμε. Να το έχετε λοιπόν κατά νου και το λακωνίζει στη φιλοσοφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, είναι σημαντικό το θέμα αυτό και οπότε θα πρέπει να ε, πω στον κύριο Κέσλερ ότι πρόκειται για πολύ σημαντική καμπή για την Ευρώπη, για τα κράτη-μέλη. Είναι θέμα επομένω εμπιστοσύνη προς ε, αυτό το θεσμό και οπότε προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια μετάβαση σε, μια σφαίρα υπερ-εθνική, υπερ-κρατική. Ε, είμαστε ταυτόχρονα φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές. Αυτός ο ένας, ο ένας μόνο εισαγγελία είναι κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί από πολιτική πλευρά ε, είναι κάτι το ξένο ω προ αυτό που ξέρουμε εμεί, αυτό που ξέρουν οι πολίτε. Αυτό δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Γιατί δεν θα έχει επαφή ουσιαστική με τα κράτη-μέλη. Οπότε θα έχει όλες τι αρμοδιότητες ενός επικεφαλής ε, κάποιας μονάδας που διεξάγει τις έρευνες. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι βουλευτές. Άρα επομένω θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες της οργάνωσης. Γιατί οι σημερινές προσπα... ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας παρέχουν εγγύησεις. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι επαφές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων σε σχέση με την πρόταση Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριε Καμέλη. Εσείς δεν θα λάβετε το λόγο. Ε, εξ αριστερών, Κέσλερ έχει κάτι συγκεκριμένο. Τελευταίος ομιλητής. Δεν έχω τη φιλοδοξία να σας απαντήσω σε ένα λεπτό, ούτε καν την απαρχή απάντησης δεν μπορώ να σας δώσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο και τους συνομιλητές ε, στο πόντιουμ, στο βήμα, αλλά και τους ε, υπόλοιπους ε, βουλευτές κτλ. Ε, μας είπατε τις ε, σκέψεις σας για το πώς εξελίσσεται η συζήτηση στην Κομισιόν. Όταν η Κομισιόν ετοιμάσει το κείμενό της, τότε αρχίζει η πραγματική συζήτηση όμως. με το Συμβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο. Μετά τις ευχαριστίες μου θέλω να σας καθησυχάσω ότι όλα τα θέματα τα οποία έχετε θέσει ήδη εξετάζονται, ήδη τα έχουμε υπόψη μας. Δεν τα ακούσατε όλα αυτά στην ομιλία μου γιατί είχα μόνο 10 λεφτά. Αλλά σας διαβεβαιώ όλους και κυρίως την κυρία όλους ότι και εγώ αλλά κυρίως η διευθύντρια η κυρία Λεμπάι έχουν εβδομαδιαίες επαφές με εισαγγελεί, με δικαστές, με εθνικές κυβερνήσεις, ακόμα και με εθνικά κοινοβούλια σε ορισμένε περιπτώσει. Σήμερα το απόγευμα μάλιστα έχω μια τέτοια ακόμα ε, συνάντηση. Θα πάω σε ένα κράτο μέλο, για να συναντήσω ε, νομομαθεί Θα συναντήσω και το Γενικό Εισαγγελία της ε, Γραφείας. Μια τελευταία διαβεβαίωση να σας δώσω που δεν έδωσα στην παρουσίασή μου και που απαντάει εν μέρη κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Ο Ευρωπαίος εισαγγελέας θα είναι 100% εισαγγελέας και οποιαδήποτε από τις δράσεις του θα υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Δηλαδή θα τον ελέγχει κάποιος δικαστής. Θα, θα ελέγχονται τα όσα κάνει ο εισαγγελέας, ο Ευρωπαίος και θα υπάρχει μια ειδική διάταξη που θα λέει ότι θα πρέπει να δοθεί άδεια από δικαστή σε περίπτωση ε, που γίνονται έρευνες οι οποίες ε, παρεμβαίνουν στα χωράφια των εθνικών δικαστών. Ε, με βάση το δίκαιο της χώρας όπου γίνεται η έρευνα και φυσικά θα εφαρμόσουμε το ουσιαστικό δίκαιο αυτό του κρατούς μέλους. Παράλληλα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ετοιμάζουν ε, μία βάση ε, για να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρμοδιότητες που θα έχει επ' αυτόν ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Τελευταία πρόταση. Ναι, σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πως πολλοί από εσάς, ειδικά από τα εθνικά κοινοβούλια, ε, έχετε κάποιες κοινέ ανησυχίες. Ε, ε, για όσους ενδιαφέρονται να το διαβάσουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια μπορούν να δουν την δήλωσή μας στο site μας ecba.org. Στη σελίδα μας λοιπόν θα βρείτε τις διευθύνσεις ε, ε, στις οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να επαναλάβω πως εκπροσωπούμε πάνω από 35 χώρες ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, οπότε μπορούμε να προσφέρουμε την εμπειρία μας στον τομέα των ποινικών υποθέσεων και θα δείτε και κάποια ζητήματα που αφορούν τη νομική πτυχή της επικουρικότητας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ λέω πρόεδρος, ε, ευχαριστώ τους ε, συμμετέχοντες, ε, τα μέλη του πάνελ, τους διερμηνείς και σερβίρεται αυτή τη στιγμή το μεσημεριανό γεύμα. Καλή σας όρεξη. Τρεις η ώρα εδώ πέρα.